Να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Ρωτώ όμω μπορούμε να ολοκληρώσουμε σε μισή ώρα για να προχωρήσουμε γρήγορα. Διότι παρατέταρτο θα έρθουν οι εκπρόσωποι της Προεδρίας. Σημείο 8 της ημερησίας διάταξης, ψηφοφορία, ο Κίσος Μπερλιγκέρ. μας εγκαταλείπει. Παρότι είμαστε η πιο ενδιαφέρουσα επιτροπή του Κοινοβουλίου. Παρά τα αυτά πρέπει να κληρώσουμε τη δουλειά σας. Αναφέρομαι στην έκθεση για τη δικασία της Μπολόνια. Θέλετε να πείτε κάτι πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ένα λεπτό έχετε. Μόνο ένα λεπτό. Θέλω να σας επισημάνω το εξής. Την παράγραφο 23 και την τελευταία τροπολογία που υπευλήθη σχετικά αργά. διότι ήταν ένα σημαντικό σημείο. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθήσω την προσοχή στην παράγραφο 23, γιατί εδώ φύγουμε το βασικό πρόβλημα της ε, όλης έκθεσης τι σημαίνει, σε τι αναφέρομαι. Η σχέση της διαδικασία της Μπολόνια, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την, την Ένωση, μάλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Το λέω αυτό γιατί στο Βουκουρέστι θα έχουμε τη διετή υπουργική διάσκεψη που θα γίνει εκτός των πλαισίων της Ένωσης. Ακούγεται περίεργο πώς ο ευρωπαϊκός χώρος της βάσης είναι εντός της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να γίνονται δραστηριότητες με κάπως περίεργο τρόπο σαν, να δίνεται η αίσθηση ότι ο ευρωπαϊκός χώρος της δοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι εκτός Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν να διευθετήσουμε στα πλαίσια της Λισαβόνας αυτό το ζήτημα. Με αυτή την τροπολογία προσπαθούμε λοιπόν να λάβουμε αυτό υπόψη και να το διευθετήσουμε. Δεν είναι λεπτομέρεια. Αυτό βασικά ήθελα να σε επισημάνω πριν την ψηφοφορία. Okay. Thank you. Ε, do you have your... Ευχαριστώ. Έχετε την κάρτα σας παρακαλώ αν χρειαστεί για την ψηφοφορία. Πάμε στην τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές Υιοθετείτε. 49. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 2. Υπέρ, κατά, αποχές Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 3, υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. «56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «57-58 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε για την 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Υιοθετείται με 12 έναντι 9. 60 υπέρ, κατά. Ξανά, για την 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές Υιοθετείτε. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές Υιοθετείτε. 69 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 70 υπέρ κατά αποχές 60, 71 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 82 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ψηφίσουμε για την 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εναντί 20 απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμό 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Υιοθετείται. Ο συμβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Υιοθετείται. Πάμε τώρα στην 100 της κυρίας Μακλάρκεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 108 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 103 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε 105 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 107 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. απόχέ 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείται. Άρα, πάμε στην 119. Στην επόμενη σελίδα. 115 υπέρ. Κατά. αποχέ, Υιοθετείτε. 124 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβασμό 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Άρα πάμε. 132 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβασμό 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Πάμε στην 141 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 141. Πέραση ψηφοφορίας. 14 10 ε, απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. και Κύριε Ναβρίδοβα, θέλετε και πάλι να ψηφίζετε, πάλι θα την απορρίπταμε. Υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα σας. Μπορείτε και πάντοτε να μου το δείχνετε με ανάταση χειρός. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Άρα προχωρούμε στην 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελεγξούμε. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 156 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για την 156 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 158 και 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχε απορρίπτεται 161 υπέρ κατά Κατά, υιοθετείται 162 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχέ, υιοθετείται 166 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχέ, υιοθετείται 165 υπέρ κατά Αποχέ. υιοθετείται 168. Πρώτο σκέλο, υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. Δεύτερο σκέλο, υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται. Συμβασμό 10, υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται. Άρα πάμε στην 169, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 173 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 174 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείτε. Γρήγορα υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε. Την 175. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 11 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Άρα πάμε στην 180. Υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 182. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 184. Υπέρ. Συγγνώμη. Λέει η Πρόεδρος. Την 184. Καταπίπτει 184. Πάμε στην 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Θέλετε έλεγχο. 201. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. πέρας 17-6 γιατί κάποιος δεν είχε ψηφίσει. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πού είμαστε. Πού. 202. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 Σιλβία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Έλεγχος για 213 άρχεται. Πέρας. 14-11. 2.14. 2.14 και 2-15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το πρώτο τμήμα της 17 Βερζιά, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Για την 11 άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. 13-12 εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 και 15 μαζί υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία 14 και 15. Πέρας. 9-17 απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά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 κατά αποχές έλεγχος. 23-1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 10-16 απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 131 ε, Μιγκάλσκι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γνωμοδότηση ΙΜΚΟ. 1. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ 15, 16 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές όλες μαζί συμπούρβουλες. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η τελική αυτή ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπερλίνγκερ. Συγχαρητήρια. ότι έκανα ένα λάθος, διότι ψήφισα αποχή. Δεν το έκανα όμως ε, εσκεμένα. Παρακαλώ να διορθωθεί στα πρακτικά. Ούτως θα γίνει. Και δεύτερο, να πω το εξή. Θέλω να ευχαριστήσω εγκάρδια όλους τους συναδέλφους, αλλά ιδίως την πρόεδρο της Επιτροπής, που ξεκίνησε αυτό το δρόμο με την έκθεσή της το 2009 καθώς αυτή την έκθεση βασίζεται και η σημερινή αυτή έκθεση. Από εκεί άντλησε την εμπνευσή μου. Και θέλω να επισημάνω επίσης το εξής. Λάβαμε μια πολύ σημαντική απόφαση και ελπίζω βεβαίως ότι θα επιβεβαιωθεί και στην Ολομέλεια. Εκφράζοντας την επιθυμία ότι η Ολομέλεια θα φτάσει στη ψηφοφορία μάλλον θα ψηφίσει το αργότερο το Μάρτιο, διότι τον Απρίλιο το ή άλλως λαμβάνει η χώρα διάσκεψη στο Βουκουρέστι, καλό θα ήταν ε, οι υπουργοί στη διασκευή του ήδη να γνωρίζουν ποια είναι η βούληση του Κοινοβουλίου. Και δεύτερο, να πω το εξή. Η σημασία της δικής μας ψήφου έγκυται στο εξή γεγονός. Έχουμε ακολουθήσει μια επικοδομητική προσέγγιση. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Εκπαίδευσης και η διαδικασία της Μπολόνια αποτελούν ένα πολύ δύσκολο και βαρύ δρόμο, δεν είναι ένας περίπατος, οπότε αν δεν υπάρξει στήριξη δεν θα γίνει τίποτα. Δεν α, μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά στη διακριτική ευχέρεια και τη βούληση των πανεπιστημίων. Γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό βασίζεται στην εθνική αρμοδιότητα. Αρμοδιότητα σημαίνει να υπάρχει έκφραση ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και αρμοδιότητα, πρέπει να υπάρχει αρμοδιότητα της Ένωσης. Μιλούμε λοιπόν για σύμπραξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν τη διαδικασία θα πρέπει να την πάμε σε απόλυτο πάθος. Ευχαριστώ. Κύριε Μπερλιγκουέρ, θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, συναδέλφους και από τις άλλες πολιτικές ομάδες να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε να έχουμε την συζήτηση για τη διαδικασία της Μπολόνια στην ε, Ολομέλεια. Δεν είναι μονάχα κάτι το οποίο ενδιαφέρει τους ε, σπουδάζοντες, Πρέπει λοιπόν όλες οι πολιτικές ομάδες και πιστεύω ότι όλες θα είναι υπέρ, να έχουμε μια έκθεση για το θέμα αυτό. Και θα πρέπει να ζητήσετε την υποστήριξη των πολιτικών σας ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ψηφοφορία τώρα. Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Έκθεση Λόκεγκαρτ. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Λόκεγκαρτ. Ωραία. Αφού δεν θέλετε, ψηφίσουμε αμέσως. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Ποχές. <clears throat> Δεκτή. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για 15. Άρχιε η ψηφοφορια περασε Πέρας. 19-6. 6-19 εν πάση απερίφθη. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 19 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία στη 19. Πέρας ψηφοφορίας. 6-17 έχασε. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή 38 κόστα υπέρ 36 υπέρ ε, έλεγχος 36. Άρχεται η ψηφοφορία στην 36. περασε 11 11-13 από την χάνη. 37 υπέρ κατά. Ορίστε. Α, εκπίπτει 37. Εντάξει, 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 <clears throat> υπέρ κατά α αποχές έλεγχος 40 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 10-14 απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 3 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 κοστα υπέρ κατά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 22 υπέρ, δύο ψηφίκατα. καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Λόκεγκαρντ. Λόγω της Δανικής Προεδρίας ερχόμαστε στην έκθεση Τούκε. Έχετε το λόγο κύριε Τούκε. για τον εξυγχρονισμό του συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Yes, thank you. I... Just a moment. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου ένα λεπτό. Tisztelt uh, kollégák, kedves Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, έχω να κάνω μια σύντομη ε, παρουσίαση. Πρόκειται για το θέμα το οποίο άπτεται των μέσων που έχουμε στην ε, Ανατολική Ευρώπη για την εκπαίδευση και είναι απαραίτητο ίσως να προτάξουμε την ε, καλύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών θεσμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση Μπορώ να σας πω ότι η διαδικασία της Μπολόνια είναι ένα τμήμα της δυσπιστίας η οποία έχει δημιουργηθεί. Ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο με απότομη, απότομα ουσιαστικά εφαρμόστηκε η διαδικασία της, της Μπολόνιας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και χώρες όπως η Ρουμανία. Αυτό λοιπόν όπως καταλαβαίνετε δεν έγινε χωρίς κάποιες τριβές οδήγησε σε αντιπαραθέσεις και σε προβλήματα στα διδακτικά προγράμματα. Και επομένως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και αυτό είναι και το αντικείμενο της εκθέσεως την οποία έχω την τιμή να παρουσιάσω και συνδέεται βέβαια με αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Μπερλίνγκορ. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δημιουργία της Μπολόνια και να εξασφαλίσουμε ότι θα ενσωματωθεί σε μια διαδικασία η οποία θα έχει και μακροχρόνια ωφέλη για τους μαθητιώντες και τις μαθητιώσεις στην τρίτο βαθμία εκπαίδευση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως μια κρίση, μια οικονομική κρίση, μια γενικότερη κρίση που αντιμετωπίζουμε να σοβεί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν ιδιαίτερα για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου τίθεται και το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για μας όχι μόνο στις δικές μας χώρες αλλά και στις χώρες της σύνολης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέχει ιδιαίτερη σημασία. Στις 20 ε, Σεπτεμβρίου του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταλήξει σε μια θέση και ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι με τον πιο ευφυή, τον πιο συμπεριληπτικό και τον πιο βιώσιμο τρόπο να εξασφαλίσουμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα στις χώρες μας. Όπως γνωρίζετε, είναι γεγονός ότι η σχολική εκπαίδευση συντελεί στη μείωση της ε, ανεργίας και φυσικά έχουμε μεγάλες δυσκολίες στον τομέα της ανεργίας σήμερα σε όλες τις χώρες μας και ξέρουμε ακριβώς πόσο σημαντική μέσα στα πλαίσια της ανεργίας είναι η ενεργεία των νέων στην Ευρώπη. Ξέρουμε <clears throat> ότι το μέσο ποσοστό της ε, ανεργίας των νέων, ακόμα και των νέων οι οποίοι έχουν υψηλά προσόντα, είναι περίπου το διπλάσιο. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν βέβαια προσόντα, είναι πολύ υψηλότερη η ανεργία των νέων. Βέβαια, παίζει κάποιο ρόλο η απόκτηση διπλωμάτων και προσόντων. Αυτοί που έχουν περισσότερα προσόντα έχουν μικρότερη ανεργία. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν προσόντα οι νέοι και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να αποφύγουν την, το φάσμα της ανεργίας. Υπάρχουν και άλλες εύγλωτες ε, στατιστικές οι οποίες μας καταδεικνύουν ότι ότι αυτή τη στιγμή μόνο 24% των εργαζομένων στην ε, αγορά εργασίας είναι νέοι με υψηλά προσόντα. Ξέρουμε ότι το μέλλον θα είναι διαφορετικό. Ξέρουμε ότι θα είναι απαραίτητο στο μέλλον, ακολουθώντας τη στρατηγική 2020, να αυξηθεί αυτό το ποσοστό να φτάσουμε το 35-40% εργαζομένων οι οποίοι θα είναι αυτοί με τα υψηλότερα προσόντα στην αγορά εργασίας. Είναι λοιπόν και μια περαιτέρω πρόκληση για μας και θα πρέπει να μας οθήσει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τρίτη τώρα στατιστική ένα τρίτο στατιστικό στοιχείο που συνηγορεί προς την κατεύθυνση αυτή είναι το γεγονός ότι μεταξύ των 500 πανεπιστημίων στον κόσμο μόνο 200 είναι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Δηλαδή τα άλλα 300 είναι σε άλλα μέρη του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε χιλιάδες πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα φαινόμενο εντυπωσιακό αυτό. το γεγονός ότι μόνο 200 από τα πανεπιστήμια μας εμπίπτουν στο χώρο της αριστείας, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και δεν είναι σχεδόν κανένα από τα πανεπιστήμια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Είναι κρανίου τόπος τα πανεπιστήμια της Κεντρικής και Ανατολικής ε, Ευρώπης. Αυτή η διαδικασία λοιπόν του εξυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και τη διαδικασία του Βερολίνου όπως αναφέρεται, ώστε να εξασφαλίσουμε την ενσωμάτωση και των πανεπιστημίων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και πιστεύω ότι όλα αυτά τα δύο προγράμματα, το πρόγραμμα της Μπολόνια που αναφέρθηκε προηγουμένως και αυτό είναι πραγματικά συμπληρωματικά. Νομίζω ότι το σύνολό τους θα μπορέσει να έχει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και είναι πολύ θετικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Κατάρτισης και Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού θέλουν, θέλει να, να εστιάσει την προσοχή της στους δύο αυτούς τομείς. Κάποιες άλλες πτυχές θα ήθελα να αναφέρω επίσης από το σχέδιο έκθεσης που έχετε όλοι στα χέρια σας, στην ε, μητρική σας γλώσσα. Εν καιρό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τροπολογίες οι οποίες θα αφορούν αυτό το σχέδιο ε, έκθεσης. Μόνο κάποιες ε, υπενθυμίσεις για την περαιτέρω εργασία μα. Είναι ρευστέ οι συνθήκε αλλάζει ο κόσμο συνεχώ. και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευελιξία και τη δυνατότητα ταχεία προσαρμογή στην εκπαίδευση. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες πανεπιστημιακής παιδείας έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό το μοντέλο το οποίο περισσότερο προωθούμε τώρα είναι το μοντέλο της διαβίου εκπαίδευσης. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτό το μοντέλο και θα πρέπει πάντα με ταχύτερους ρυθμούς να εξασφαλίσουμε την ε, περαιτέρω και διαβίου εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παροτρύνουμε τους διδάσκοντες και τους ε, σπουδάζοντες να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα και να την ε, προωθήσουμε και στο εσωτερικό αλλά και μεταξύ κρατών μελών. <clears throat> Να υπάρξει λοιπόν διαπερατότητα μεταξύ χωρών και μεταξύ τομέων του επιστητού. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη σημασία ε, στο να υπερπηδήσουμε, να ξεπεράσουμε και το εικονικό κατά κάποιο τρόπο σιδηρούν παραπέτασμα που υπάρχει λόγω της μεγάλης διαφοράς στα επίπεδα εκπαίδευσης στην Ανατολική και την Δυτική Ευρώπη. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα τα πανεπιστήμια στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη υποστήριξη. Λόγω λοιπόν αυτού του γενικού πλαισίου θα είναι απαραίτητο να κάνουμε και τις απαραίτητες επενδύσεις και να προωθήσουμε και καινοτόμες μεθόδους διδαχής. Κοστίζουν όλα αυτά, αλλά μπορεί να πει κανείς και η δημοκρατία κοστίζει. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η γνώση θα υποστηριχθεί γιατί η γνώση είναι μία από τις βάσεις της κοινωνίας μας και επομένως είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις ιδίως στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Όλες αυτές οι επενδύσεις έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και αποδίδουν τα μάλα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Αν ατενίσουμε την αγορά εργασίας και δούμε ποια είναι η σχέση της αγοράς με τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές σπουδές, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο αυτών κόσμων. Πρέπει αυτό το χάσμα να μειωθεί στο μέλλον. Και στόχος αυτής της έκθεσης είναι να συμβάλλει στο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να μπορέσουμε να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και του κόσμου της αγοράς. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει και παρακολούθηση των ακαδημαϊκών για να είναι φανερό πόσο λειτουργούν για τον χώρο της ε, αγοράς. Στην εποχή του Τσαουσέσκου είχε ιδρυθεί ένα πανεπιστήμιο στη Ρουμανία, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, το οποίο στη συνέχεια μπόρεσε να αποκτήσει την πλήρη πιστοποίηση. Για τη δική μας περιοχή λοιπόν στην Ρουμανία ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε με τις εργασίες αυτού του πανεπιστημίου να παρακολουθούμε καλύτερα την κατάσταση της εργασιακής αγοράς, να παρακολουθούμε κατά πόσο υπάρχουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και να δίνουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις και στους αποφύτους. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρξαν τομείς νευραλικοί όπου οι απόφοιτοι μας μπορούσαν να βρουν αμέσως τέσσερις εργασίες, ενώ αλλού ήταν πολύ δύσκολο. Επομένως, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ αγοράς και πανεπιστημίου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το θέμα της καλύτερης συνεργασίας με εξωτερικούς εταίρους. Ο πανεπιστημιακός κόσμος λοιπόν θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην ε, ε, τοπική κοινωνία με τις εταιρείε, με τις ε, οργανώσεις κοινωνίας του πολιτών. Ιδίω λοιπόν αυτό είναι απαραίτητο σε χώρες που έχουν προβλήματα και είναι απαραίτητο και στα πλαίσια της οικονομικής δραστηριότητας να προετοιμάζεται κόσμος ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το επίπεδο. Κάναμε και συμφωνίες με την Ουγγρική ε, κοινότητα στην Ρουμανία ώστε να μπορούμε να προετοιμάσουμε και αποφύτους οι οποίοι μπορούν να εργαστούν και στις δύο αυτές γλώσσες. Ανεφέρθηκα ήδη στην έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των κρατών μελών στα θέματα της ε, ε, εκπαίδευσης. Η δική μου περιοχή βρίσκεται στα σύνορα <clears throat> μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας και η Ντέμπρετσαν και η Οραντά βρίσκονται στις δύο ε, πλευρές των σύνορων αλλά υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ αυτών των περιοχών όπως και της περιοχής του Σέγκετ και του ε, Τέμεσβάρ και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι συνεργάζονται τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων μας. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει επίσης όμως να γίνει πραγματικότητα μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Κεντροανατολικής Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε <clears throat> να καταλήξουμε και σε κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, να υπάρξει, παραδείγματος χάρη για μας είναι απαραίτητο να έχουμε ένα κοινό επίπεδο στην ε, διδαχή της ουγγρικής ε, ε, γλώσσας με κοινά σχέδια ε, διδαχής για να εξασφαλίζεται ισόρροπο επίπεδο γνώσης και στην ρουμανική πλευρά και στην ουγγρική πλευρά. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την κινητικότητα των διδασκόντων και των διδασκομένων. Ο έρασμος είναι μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας ήταν ένα από τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 10.000 φοιτητές είχαν μέχρι στιγμή την ευκαιρία να <clears throat> σπουδάσουν σε μια άλλη χώρα και θα κλείσω εδώ ένας ε, ανιψιός μου ένας εγγόνος μου μάλλον μπορούσε να, να εργαστεί στην ε, Γαλλία και μετά να ξαναγυρίσει στην ε, στη Ρουμανία. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε την επανενσωμάτωση αυτών των ε, αποφύτων οι οποίοι έχουν υψηλά προσόντα και έτσι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ολοκλήρωση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απαραίτητο με καλύτερες επενδύσεις να εξασφαλίσουμε αυτή την εναρμόνιση ιδίω στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών και να κάνουμε τι απαραίτητε επενδύσει. Τα χρήματα βέβαια είναι απαραίτητα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια περίοδο λιτότητα σε σχέση με τον προπολογισμό τη. Είναι κατανοητό αυτό, αλλά θα ήθελα να σα ζητήσω να μην κάνουμε περικοπές στον τομέα τη εκπαίδευση. Και θέλω να παρακαλέσω και την Κομισιόν να λάβει αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος έχετε καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα σε σχέση με την ε, ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μονάχα <clears throat> στα πανεπιστήμια της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με τη διαδικασία της Μπολόνιας. Όλοι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και έχετε και ένα πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων, γιατί το δικό σας σύστημα ούτως ή άλλως μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου έπρεπε να τροποποιηθεί. Για μας ήταν πολύ δύσκολο να πείσουμε τα πανεπιστήμια ότι πρέπει να αλλάξουν την διαδικασία τους. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά τα οποία μας είπατε, για την κατάσταση στην Ρουμανία και την διαμεθοριακή προοπτική συνεργασία μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε πέντε ε, βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι γιατί είναι πρώτον πυλών η Ιδανική Προεδρία. Θα ήθελα μέχρι τις 10 η ώρα να τελειώσει αυτή η συζήτηση και θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε. Κύριε Βινταλόγα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπε ο εισηγητής. Πρόκειται για μια καλή βάση ε, μόνο μερικέ τροπολογίε θα χρειαστούν για να βελτιωθεί περαιτέρω. Εγώ όμως συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Πράγματι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ ε, Ανατολικής και, Ευρω... και Δυτικής Ευρώπης. Και εσείς προτείνετε ένα ε, πρότυπο συνεργασία σε βάση των κύκλου σπουδών. Είναι μια καλή βάση αυτή, πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο σύστημα ε, που μπορούν να αξιοποιήσουν ε, οι φοιτητέ και οι απόφοιτοι. Άλλο σημαντικό στοιχείο, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Το στερίζουμε και αυτό το στοιχείο γιατί αυτό θα μας ε, βοηθήσει να καθορίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται οι αποφοιτοί μας. Για παράδειγμα, τις γλώσσες που πρέπει να γνωρίζουν. Να τους υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να στραφούν και προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι δεν πρέπει να παράγουμε μόνο από φύτους και εργαζομένους, αλλά πάντα να έχουμε κατά νου και την ε, δημιουργία νέων αξιών. Όχι δηλαδή μόνο ε, να έχουμε ένα προϊόν για την αγορά εργασία, να θυμόμαστε ότι ε, βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους να αναπτυχθούν περαιτέρω. Αναφερθήκατε στη σημασία αυτής της μετάβασης από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αποφύτους σε αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό και για μας, ως μέλη του Κοινοβουλίου, να είμαστε σε θέση να εκφέρουμε γνώμη ε, για, τη, για αυτά τα συστήματα κατάρτισης. Και εμείς έχουμε εδώ πέρα ασκούμενους οι οποίοι δεν ε, αμείβονται. Και αν θέλουμε καλές ε, συνθήκες εργασίας, από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέμπ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τόκας και να το συγχαρώ για την ενδελεχέστατη ανάλυση του σε σχέση με, την, ε, με τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας της ε, Μπολόνια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι το τρίτο ή τέταρτο έγγραφο το οποίο αντιμετωπίζουμε για τα θέματα αυτά. Θέλω να σας υπενθυμίσω <clears throat> την εξαιρετική έκθεση του κυρίου Σμιτ σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Εγώ ο ίδιος εκπώνησα μια έκθεση για τους νέους και για την κινητικότητα. Υπήρξε η έκθεση του κυρίου Μπερλιγκουέρ για τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της διαδικασίας της Μπολόνια. Και εδώ έχουμε μια έκθεση η οποία αφορά περισσότερο την εσωτερική δομή της, ε, του εξυγχρονισμού των πανεπιστημίων. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μέσα σε αυτή τη θητεία ξεκινούμε να εξετάσουμε από την αρχή όλη τη διαδικασία της Πολώνιας. Χρειαζόμαστε μια πολιτική συνένεση για να δώσουμε το κατάλληλο πολιτικό μήνυμα σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει το παλιωμοδίτικο πανεπιστήμιο, η παλιά δομή στα πανεπιστήμια, που αποτέλεσε και εμπόδιο για την ε, συνέχιση και την εμβάθυνση της διαδικασίας της Μπολόνια, που είναι όμως μια πολύ σημαντική διαδικασία. Στην ε, Δυτική Ευρώπη βέβαια υπήρξε μια μεγαλύτερη πρόοδος, αλλά οι χώρες οι οποίες είχαν βρεθεί στο κομμουνιστικό στρατόπεδο στο παρελθόν είναι αυτές για τις οποίες η διαδικασία της Μπολόνια είναι και η πιο σημαντική. Θυμάμαι την εποχή της δημοκρατικής μετάβασης. Υπήρξε το θέμα της αυτονομίας των πανεπιστημίων, δεν υπήρξε η απαραίτητη μεταρρύθμιση στα θέματα αυτά Γι' αυτό θα πρέπει να καλυφθεί και το υπόλοιπο τμήμα της μεταρρύθμισης και να προωθηθεί η διαδικασία της Μπολόνιας και αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν προβλήματα μονάχα στην Δυτική ή στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ευρώπη σαν σύνολο, σαν Ήπειρος θα πρέπει να επιταχύνει την διαδικασία της Μπολόνια εάν θέλουμε πράγματι στα σοβαρά να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικά τα πανεπιστήμια μας εναντί αυτών της Ανατολικής Ασίας και του αγγλοσαξονικού κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Λάσλο κάλυψε πολλά στοιχεία. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Έκανε ορισμένες εξαιρετικές παρατηρήσεις που θα πρέπει να εξελίξουμε περαιτέρω τουλάχιστον εδώ και να δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες, ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια, για να ακολουθήσουν το ρυθμό της ε, κοινωνίας και του ορίζοντα 2020 με τους στόχους που έχουμε θέσει. Γιατί σίγουρα όλα αυτά αποτελούν, είναι στοιχεία κέρια σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Αν δεν ε, τα καταφέρουμε, τότε οι νέοι εργαζόμενοι δεν θα έχουν ε, τι απαραίτητες δεξιότητες και δεν θα είναι ανταγωνιστική Ευρώπη. Αυτό το στοιχείο που από τα 200 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από τα 500 ε, καλύτερα του κόσμου, εντάξει δεν είναι και πολύ άσχημα αλλά δεν είναι ικανοποιητικό. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι σε ορισμένα πανεπιστήμια ε, τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα από ό,τι σε άλλα και από εκεί μπορούμε να αντιλήσουμε ένα μάθημα. Ορισμένοι από του εκπροσώπου, καλό μάλλον θα ήταν να καλέσουμε ορισμένου από του εκπροσώπου των ε, καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου και να του ε, πάμε στα λιγότερο καλά. Ε, και πλέον δεν ισχύει αυτό που λέγαμε παλιότερα ότι πρόκειται για ανεξάρτητα κράτη που πρέπει να καθορίσουν μόνο τους το σύστημά τους. Πέρυσι είχαμε πάει στο Σεντιάκο, το Κοποστέλα και εκεί πέρα είδαμε αυτό το παράδειγμα της ε, ε, καινοτομίας ε, που απαιτείται. Αντί δηλαδή να κρίνουμε τα πανεπιστήμια από τον αριθμό των δημοσιεύσεών τους, καλύτερα θα ήταν να ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση, γιατί οι δημοσιεύσεις δεν είναι απαραίτητα και το κατάλληλο κριτήριο. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα πανεπιστήμια μας θα ακολουθούν τα κριτήρια που έχουμε, καλέ, θέσει. Είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τέλει. Παλιαδέλη. Ναι, καλή σας μέρα. Ε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι η Επιτροπή ασχολείται τόσο έντονα το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ε, αυτό προκύπτει και από την ανάγκη για την ανανέωση ε, των πανεπιστημιακών σπουδών ε, και από την ανάγκη για την αγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον ε, συνάδελφο κύριο Τόκες για, το, για τη δουλειά του, όπως και τον κύριο Μπερλίνγκερ για τη δική του και να κάνω πολύ σύντομα μερικέ παρατηρήσεις οι οποίες δημιουργούν κάποια ζητήματα. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση σε παγκόσμιο επίπεδο των πανεπιστημίων υπάρχουν ήδη δημοσιευμένες αμφισβητήσεις για τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση. Επομένως, ε, ίσως μια απάντηση της ευρωπαϊκής ε, κουλτούρας θα ήταν να δημιουργήσει ένα δικό της σύστημα αξιολόγησης, να προτείνει αυτή ένα δικό της σύστημα αξιολόγησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν αξίες ή τρόποι διδασκαλίας ή standards στα οποία τα πανεπιστήμια της Ευρώπης θα είχαν ενδεχομένως και τα άλλα πανεπιστήμια στον κόσμο θα έπρεπε να ξαναδούν και εκείνα τα προγράμματα σπουδών τους. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι του Χονγκ Κονγκ και η Σανκάη είναι οι απόλυτοι κριτές ε, με βάση, ε, τα, κριτήρια των οποίων θα πρέπει να προσαρμοστούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έχουμε μια παράδοση στη γνώση που θα έπρεπε να την αξιοποιήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, θεωρώ επίσης ότι υπάρχουν μερικοί όροι στην, ε, στο, στην φρασιολογία που χρησιμοποιούμε στα κείμενα και στις προσκλήσεις για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επίσης είναι παραπλανητική για αρκετά πανεπιστήμια της ε, Υπήρου μας. Όπως για παράδειγμα η ε, Innovation που θεωρώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, σημαίνει πράγματα τα οποία ορισμένες τάσεις δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τίποτα και υπάρχουν τέτοιοι κλάδοι που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την επιστήμη τους με βάση τη λογική της πρωτοποριακής προσέγγισης. Αυτό δεν σημαίνει μη διεπιστημονικότητα, αλλά οπωσδήποτε το innovation δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μία άλλη αγκύλωση που θα έπρεπε ίσως να την εξετάσουμε με αυτή την αφορμή είναι η όρος έρευνα που σχεδόν πώς να πω, αποκλειστικά παραπέμπει σε εργαστήρια χημίας, ιατρικής, φαρμακευτικής κλπ. Ούτε αυτό νομίζω ότι είναι σωστό γιατί η έρευνα τουλάχιστον στην Ευρώπη θα έπρεπε να ε, διευρύνεται και σε άλλους κλάδους ε, που δεν είναι αναγκαστικά δεμένοι με την, μόνο με την εργαστηριακή έρευνα. Και μια παρατήρηση που αφορά στην ανεργία των παιδιών που δεν έχουν πάει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προέρχομαι από μια χώρα που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί πτυχιούχοι χωρίς ε, εργασία και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης και όχι ε, ο αριθμός των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τελειώσω με μια πολύ επικίνδυνη κατά την εκτίμησή μου σύνδεση του των προγραμμάτων σπουδών με τις επιχειρήσεις. Είναι βεβαίως πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για την ε, απασχολησιμότητα των πτυχιούχων μας ε, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Όμως έχει παρατηρηθεί το γεγονός και έχουν δημοσιευτεί επίσης ζητήματα που αφορούν στην προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών με βάση τα αιτούμενα των επιχειρήσεων. Αναρωτιέμαι αν σε ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα ήταν σκόπιμο να ακολουθούμε τις προδιαγραφές που μας δίνει μια ιδιωτική επιχείρηση προκειμένου να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα σπουδών μας. Είναι ένα επικίνδυνο σημείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Συμφωνώ ωστόσο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και την διαδικασία της Μπολόνια, να τη διευρύνουμε, και την διαδικασία της αξιολόγησης και την διαδικασία προσαρμογής σε μοντέλα τα οποία θα επιτρέψουν στους πτυχιούχους των μελών κρατών να εργαστούν και να απασχοληθούν σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνατε κύριε Τόκες. Κύριε Σέβερτ, κύριε Έβερτ, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Τόκες. Μόνο μία υπενθύμηση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ότι όλες αυτές οι εκθέσεις που έχουμε εγκρίνει με μεγάλη πλειοψηφία όπως του κυρίου Μπελιγκουέρ και η δική σας έκθεση να μην, ε, ε, να μην καταλήγουν σε αντιφάσεις, να έχουν μια ενιαία γραμμή. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητη μια καλή πανεπιστημιακή παιδεία η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την τωρινή κρίση. Δεν σημαίνει αυτό ότι από τη στιγμή που έχουμε ξεπεράσει την κρίση θα μπορούμε να παραγνωρίσουμε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η καλή εκπαίδευση και η έρευνα και η κατάρτιση είναι μόνιμες αξίες και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε μόνιμο επίπεδο υπάρχει η κατάλληλη διαδικασία. Εγώ πάντα έχω και ένα πρόβλημα με την, το σημείο 5 της ε, έκθεσής σας, το οποίο αναφέρεται στην στάση που θα πρέπει να κρατήσει η Κομισιόν σε σχέση με, το, με την κατάταξη των ε, Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Εγώ νομίζω ότι μια κατάρτιση, μια, κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ευρώπη δεν είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε αντίθετα είναι να μπορούμε να πληροφορήσουμε <clears throat> τους φοιτητέ και τους, επό... τους φοιτητέ οι οποίοι θα έρθουν στο μέλλον ποιες είναι οι δυνατότητες οι οποίες έχουν για να σπουδάσουν για κάθε συγκεκριμένο τομέα. Αλλά μια κατάταξη δεν νομίζω θα βοηθήσει. Ναι, πέτρα το σημείο 5. Δεν είναι, περιλαμβάνει μονάχα την κατάταξη, αλλά έχει μια ευρύτερη ε, διατύπωση. Τονίζει την ανάγκη να υπάρξει και καλύτερη ποιότητα των ε, διδασκάλων κτλ. Ο κ. Παπα-Νικολάου τώρα. Ε, I also want to thank Mr. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τόκες για την ολοκληρωμένη του αυτή η έκθεση. Συμφωνώ απολύτω με την ανάγκη να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό μας, στα εκπαιδευτικά μας συστήματα και στην ε, ε, γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εκπαίδευσης και της αγορά εργασίας. Θα ήθελα να προσθέσω ε, κάτι στα όσα είπε η κυρία Παλιαδέλη. Κανένας δεν λέει ότι πρέπει να ακολουθούμε τις αγορές, τις απαιτήσει δηλαδή της αγοράς. Αυτό που λέμε είναι σημαντικό για ένα κράτος μέλος της Ευρώπης να ξέρει ότι τα επόμενα χρόνια, για παράδειγμα, θέλουμε πολλούς εργαζομένους στον τομέα της πληροφορικής και έχουμε πάρα πολλούς δικηγόρους, για παράδειγμα, όπως είμαι εγώ. Κανένα δεν διαφωνεί λοιπόν με αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω. Λέμε στη στρατηγική μας ε, για το 2020 ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στο τρίγωνο της και ε, εκπαίδευση, καινοτομία, έρευνα. Και εμείς συμφωνούμε. Πώς να συμφωνήσουμε πρέπει να συμφωνήσουμε μάλλον, πώς να συμφωνήσουμε με όλα όσα υπό, υπόθηκαν εδώ στην Επιτροπή μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ε, εθνικό επίπεδο παράλληλα να έχουμε αποτελεσματική χρηματοδότηση. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε εν μέσω μιας τέτοιας κρίσης να συνεχίσουμε με μείωση του υπερπολογισμού για την παιδεία σε πολλές από τις χώρες μας στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται για κάθε κράτος μέλος και σε πολλά από αυτά τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα για όσα βρίσκονται σε περίοδο μεγάλης ύφεση και έχουν μεγαλύτερα προβλήματα σχέση με άλλα κράτη-μέλη, έχουν, πολύ, έχουν κάνει πολύ σημαντικές περικοπές ε, στα, στη χρηματοδότηση της παιδείας. Μπορούμε λοιπόν σε αυτή την έκθεση να προσθέσουμε ένα σχόλιο ότι δηλαδή καταδικάζουμε αυτή την προσέγγιση, αν συμφωνεί βεβαίως και ο εισηγητής. Θα μπορώ να το αποστείλω ένα σημείωμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε εδώ, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ. please, the next three I have... Ευχαριστώ. Οι επόμενοι ομιλητέ θα είναι πάρα πολύ σύντομε, γιατί μα περιμένουν οι Δανείοι. κύριε Μπόρις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του και να πω ότι το γεγονός και μόνο ότι εστιάζεται στην ποιότητα ε, της εκπαίδευσης, αυτό είναι το σημαντικό. Ακόμα και σε εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση και η επένδυση στην παιδεία θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ποιότητα. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνω το γεγονός ότι και οι τέχνες ε, έχουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ε, παιδείας. Τα τα ταμεία και όλα τα σχετικά κονδύλια της Ένωσης θα πρέπει να χρηματοδοτούν με βάση την ποιότητα. Ευχαριστούμε για την ε, συντομία κύριε Σβάλτσκι. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την έκθεση κύριε Τόκης. Και εγώ ανήκω στον ακαδημαϊκό κόσμο, οπότε πραγματικά το θέμα που αγγίζεται είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και εγώ είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να δώσουμε το βάρος στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Ο αριθμός των σπουδαστών δεν μεταφράζεται αναγκαστικά σε ποιότητα. Πολύ συχνά βλέπουμε στην Πολωνία να έχουμε στρατιές ανέργων πτυχιούχων. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια αντίστοιξη ανάμεσα στον ακαδημαϊκό κόσμο και τις υψηλές δεξιότητες. Οι υψηλές δεξιότητες θα πρέπει να προσφέρουν θέσεις εργασίας, ενώ ε, το πανεπιστήμιο ως πανεπιστήμιο προσφέρει και πρέπει να προσφέρει εκπαίδευση, παιδεία, γνώση. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο δεν έχει ως μοναδικό σκοπό την προετοιμασία των εργαζόμενων για την αγορά εργασίας. Δεν θα πρέπει να σκοτώσουμε, αν θέλετε, αυτή την βασική, το βασικό χαρακτηριστικό των πανεπιστημίων. Όσον αφορά τώρα τη νέα κατάταξη των πανεπιστημίων, θα έλεγα ότι αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο των ευρωπαϊκών ανώτατων ιδρυμάτων, η λύση δεν είναι η κατάταξή τους, ε, η βαθμολογία τους αν θέλετε και η διαβάθμιση τους. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι η λύση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αυτονομία των πανεπιστημίων, όπως και την αυτονομία των κρατών μελών για τη χάρεξη του συστήματος παιδείας τους. Ευχαριστώ θα αναφερθώ, μάλλον θα ανακοινώσω μόνο τα σημεία στα οποία θα αναφερθώ αργότερα με τροπολογίε. Πρώτα απ' όλα, το θέμα τη κατάταξη των πανεπιστημίων. Ουσιαστικά, εμείς είμαστε Υποτελεί στα αγγλικά, μάλλον πανεπιστήμια, τα 200-500 πανεπιστήμια που λέμε, ε, ουσιαστικά ε, σε τι μεταφράζονται. Επ' αυτού λοιπόν συμφωνώ πολύ με τη συνάδελφο την κυρία Παλιαδέλη. Δεύτερο, κάτι σημαντικό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην προσπάθεια ενοποίησης προγραμμάτων σπουδών και ε, ισοτιμίας ε, τίτλων σπουδών, δηλαδή ένα μηχανικός, ένας γιατρός που μπορεί να εργαστεί και στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα, ναι, θα πρέπει εκεί να υπάρχουν ευρωπαϊκά κριτήρια. Από την άλλη όμω, η ιδιαιτερότητα των ανθρωπιστικών σπουδών ε, θα πρέπει να διαφυλαχθεί από την άλλη θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυστηροί σε ό,τι αφορά την επαγγελματική προετοιμασία του καθενός, γιατί εκεί εξαρτάται, αν θέλετε, και η ζωή του ανθρώπου, αν θέλετε, σε πολλά επαγγέλματα, και να αφήσουμε τις τοπικές κουλτούρες και συμπεριφορές να ε, υπάρχουν, γιατί αυτό είναι ένας μεγάλος πλούτος. Και σίγουρα μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι σε ό,τι αφορά τα διάφορα επαγγέλματα, οι σχετικέ σχολέ που προετοιμάζουν επαγγελματίε να έχουν, αν θέλετε, και μια συνιστόσα, ε, μια διάσταση ανθρωπιστικών σπουδών. Ιδάλω προετοιμάζουμε μόνο ρομπότ για να βγουν να ασκήσουν ένα επάγγελμα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ναι, κατάλαβα, Πρόεδρε. Εντάξει, τα υπόλοιπα αργότερα. Μπορεί να γίνει με τροπολογίες. Ναι, η κόμιση, κύριε Τάισον, δύο λεπτά ή δυνατόν. Και λιγότερο, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσα ακούστηκαν σήμερα και μπορούμε να στηρίξουμε ε, σε μεγάλο βαθμό το κείμενο όσο έχει αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε τον Τόκες για την προσπάθειά του. Λίγα σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσα υπόθεσαν για την ποιότητα και την συνάφεια της εκπαίδευσης. Ε, είναι πολύ σημαντικό οι σπουδαστέ να έχουν τι κατάλληλε δεξιότητε για να μπορούν να συμμετοχθούν στο αγορά εργασία γρήγορα. Και αν η ποιότητα αυξάνει, τότε οι τυχιούχοι είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλου εργαζόμενου στην αγορά εργασία. Κυρία Πρόεδρε, επίση, εσεί απαντήσατε ε, στο θέμα τη κατάταξη των πανεπιστημίων είναι κάτι που το στηρίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Και το σύστημα κατάταξη το σχεδιάζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Και θέλω να επανέλθω και εγώ στο θέμα των πανεπιστήμιων στη Δυτική Ευρώπη και στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Φυσικά υπάρχουν διαφορέ και προκλήσει και γι' αυτό υπάρχουν τα δεκαταμία. Και να μην ξεχνάμε ότι 80 δισεκατομμύρια ευρώ από την ταμεία δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί από τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και θα μπορούσαν να συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην ποιότητα σε το βάθμιο εκπαίδευση. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν. 2 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου λοιπόν πρέπει να καταθέσετε τις τροπολογίες. Το υπενθυμίσω. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δείχνει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα τη πανεπιστημιακής εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ερχόμαστε <clears throat> στο σημείο 10 τη ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να υποδεχθώ την, κυρία Κριστίνα Αντορίνη που είναι ε, Υπουργός για την Παιδεία και την Παιδική Ηλικία τη Δανίας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και ελπίζουμε θα μας δώσετε και νέα ενάψματα για περαιτέρω πρόοδο στην επόμενη, στους επόμενους έξι μήνες στα θέματα αυτά της παιδείας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ, κυρία Πρόεδρε, όπως και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής σας. Είναι χαρά για μένα να είμαι σήμερα μαζί σας και να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο ε, Παιδείας και Νεολαίας. Εγώ ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο ε, παιδείας ε, και νεολαίας ε, πέρυσι τον Οκτώβρη και προσβλέπω πραγματικά συζήτηση που θα έχουμε και αργότερα. Να πω ότι η Δανία πρώτα απ' όλα είναι ένα μέρος του τρίου των Προεδριών με Πολωνία και Κύπρο και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με αυτές τις δύο χώρες όπως και με τις υπόλοιπε χώρες στο Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα κατάλληλα θεμέλια για να μπορούμε να συνεχίζουμε να οικοδομούμε σε αυτά για να έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η η Προεδρία επίτυχε, ε, επέτυχε σημαντικά αποτελέσματα και εμείς ξεκινούμε από εκεί που σταμάτησε η Πολωνική Προεδρία. Και αυτό αφορά και την πρόταση ε, για το Εράσμους για όλους που θα ε, θέσω σε λίγο. Να πω ότι η Δανία ανέλαβε την Προεδρία στο Συμβούλιο μια χρονική στιγμή πολύ δύσκολη, καθώς τα φώτα, αν θέλετε, πέφτουν πάνω στο ζήτημα της οικονομικής κρίσης. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια και τιτάνια προσπάθεια, αν θέλετε, για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ιδίω αυτό αφορά τους νέους. Όταν μιλούμε για τους νέους και την εκπαίδευση, να πω ότι αυτό θα είναι κάτι που θα απασχολήσει πάρα πολύ τη Δανική Προεδρία με μια σειρά πρωτοβουλειών ώστε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των νέων τουλάχιστον για την εξέβρεση μιας ε, ε, εργασίας. Γι' αυτό θα οργανώσουμε μια σειρά ε, διασκέψεων και λοιπόν εκδηλώσεων την Άνοιξη ώστε να συζητήσουμε τα θέματα της παιδείας, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και την εξέβρεση των εργασίας για τους νέους το Συμβούλιο θα διοργανώσει ε, τις ε, δηλώσεις αυτές με πρωτοβουλίες Δανικής Προεδρίας ε, που στο κέντρο θα είναι η απασχολησιμότητα των νέων και θα εξετάσουμε μεταξύ άλλων πώς η παιδεία μπορεί να συμβάλλει στα πλαίσια στρατηγικής του 2020 ώστε να έχουμε περισσότερες και καλύτερες εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την παιδεία. Θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν νωρί το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό να φτάνει το μέγιστο 10% και να αυξήσουμε κατά 40% τουλάχιστον τους νέους ε, που ξεκινούν την τετοβάθμια εκπαίδευση. Να πω ότι οθετήθηκε πρόσφατα η κοινή έκθεση για τη στρατηγική πλαίσιο 2020 ε, το υπονομαζόμενο ET 2020. Το σχέδιο αυτής της έκθεσης ε, περιέχει πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν μια καλύτερη διάδραση ανάμεσα στο ET 2020 και την Ευρώπη 2020. στόχος είναι όλες οι πρωτοβουλίες από των οποίων εργαζόμαστε να χρησιμοποιηθούν ένα κατάλληλα εργαλεία για να μας, μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους συνολικούς ε, στόχους της στρατηγικής 2020. Εν προκειμένου, η παιδεία θεωρούμε ότι έχει κομβικό ρόλο και η έκθεση ET 2020 ε, έχει μία σειρά προτεραιοτήτων να αναθέσει και μεταξύ αυτών είναι η μείωση των ε, νέων που εγκαταλείπουν νωρίς ε, την εκπαίδευση, ενίσχυση της διαβίου μάθησης και ενίσχυση της κινητικότητας. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτό αυτά τα θέματα, καθώ είναι κοινέ προκλήσει για όλου. Το βασικότερο καθήκον για την Ιδανική Προεδρία είναι διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το Εράσμου για όλου. Θα γνωρίζετε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την νεολαία, που περιέχει και ένα κεφάλαιο για τον αθλητισμό. Η Επιτροπή προτείνει μια σημαντική αύξηση σχετικού προπολογισμού κατά 70%. Και αυτό φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή αντιμετωπίζει πλέον ε, την παιδεία ε, πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να ξέρουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στην απολυσχολησιμότητα και την παιδεία και ταυτόχρονα αναγνωρίζοντα ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσχερή οικονομική κατάσταση που μα αναγκάζει να κινούμαστε πολύ περιοριστικά. Ο προπολογισμό βεβαίω ε, θα είναι το αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσια ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που αυτή τη στιγμή συζητείται στο Συμβούλιο. Ήδη αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει πλέον επισήμως κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Η Επίτροπος, η κυρία Βασιλείου, από ό,τι ε, γνωρίζω, έκανε μια σχετική παρουσία στους προηγουμένους μήνες στην Επιτροπή σας και η συνιστόσα της νεολαίας και των ανεπίσημων μορφών εκπαίδευσης είναι κάποια από τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι θα είναι και κομβικά στοιχεία και στην πραγματεύση στο Συμβούλιο. Είναι πολύ ε, σημαντική πρόκληση να θέσουμε την νεολαία ε, στο κέντρο αυτών των πρωτοβουλειών και επίσης ε, ένα, μια άλλη βασική πρόκληση είναι η παιδεία για όλους, όλες τις ηλικίε. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι ακόμα και το ίδιο το όνομα, ε, βεβαίως, ε, Εράσμους για όλους, είναι κάτι που έχει δημιουργήσει πολλά σχόλια. Πρέπει σε κάθε πρωτοβουλία να υπάρχει και ένα όνομα. Αν κάποιοι συμφωνούν περισσότερο ή λιγότερο, είναι και αυτό θεμητό, αλλά αν θέλετε δευτερεύουν προ... μάλλον φιλοδοξία της Δανικής ε, Προεδρίας είναι στο Ερεινό Συμβούλιο να έχουμε μία κάποια συμφωνία, τουλάχιστον για το περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, αυτό είναι αρμοδιότητα των Υπουργών Οικονομικών. Αν θέλουμε να ταποκριθούμε στις προσδοκίες ε, που έχουμε θέσει, θα πρέπει να εστιάσουμε ε, στην προετοιμασία του Συμβούλου Υπουργών. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις όπως σας είπα, ξεκίνησαν πλέον στο Συμβούλιο. Θα έχουμε συνεχείς επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη των πραγματεύσεων για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία σε όλα αυτά τα project. Εμείς προσβλέπουμε συνεργασία με τον εισηγητή σας όταν ορίσετε εισηγητή για αυτό το θέμα. Κάποιο άλλο σημαντικό θέμα για την Προεδρία μας είναι η διαπραγμάτευση κάποιων κριτηρίων, κάποιων benchmarks για την επιλεξιμότητα στην απασχόληση. Το 2009 κλείθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια σχετική πρόταση για τα benchmarks για την επιλεξιμότητα στην απασχόληση και την κινητικότητα και υιοθετήθηκαν πρόσφατα τα σχετικά benchmarks για την κινητικότητα. Ελπίζουμε λοιπόν στο Συμβούλιο Υπουργών του Μαΐου να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και τα σχετικά benchmarks για την επιλεξιμότητα στην απασχόληση. Φυσικά αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε κάποια τέτοια benchmarks. Πώς μπορεί κανείς να ορίσει αυτά τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα στην απασχόληση, με βάση βεβαίως την ποιότητα της παιδείας, της εκπαίδευση, Φυσικά σημαντικό ρόλο προκειμένου παίζει και η οικονομική ε, συγκυρία αλλά και η κατάσταση της αγοράς εργασίας εν γέννη. Η υιοθέτηση αυτών των benchmarks θα είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι δηλαδή η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί στην απασχόληση, στην εργασία. Δυστυχώς το επίπεδο της ενεργείας μεταξύ των νέων είναι πάρα πολύ ανησυχητικό Βεβαίω, συμφωνούμε ότι η παιδεία και η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται στην απασχόληση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η δυνατότητα ε, των πολιτών ε, να έχουν πρόσβαση στην παιδεία είναι κάτι γενικότερο, μια γενικότερη αξία και είναι ένα κομμάτι της ε, γαλούχησης του ίδιου του πολίτη. Να πω ότι στο Συμβούλιο επίσης δουλεύουμε και μία πρόταση για την αναγνώριση των προσωπικών, των ατομικών προσώτων και δεξιοτήτων. Θεωρούμε ότι και αυτό ο τομέα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τον ενισχύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πω το 2006 δεν έχει γίνει τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν υιοθετήθηκε μια απόφαση για την αναγνώριση των προσωπικών δεξιοτήτων στον ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτά τα ατομικά προσόντα δεξιότητε είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε εργαζόμενο περιμένουμε μια σχετική πρόταση Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής ε, που πιστεύουμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή την Άνοιξη. Δεν φιλοδοξούμε να ολοκληρώσουμε βεβαίω τη συζήτηση και την υιοθέτηση πρόταση αυτή κατά τη Προεδρία μα, αλλά πιστεύουμε ότι σύντομα θα μπορέσει το Συμβούλιο να υιοθετήσει ένα σχετικό ψήφισμα. Πώς ακούσατε και από τη δική μου δήλωση, Πιστεύω ότι κατανοείται ότι η νεολαία για μας ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμά μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας μελλοντικέ γενιές και οι στόχοι της απασχολησιμότητας και της ανάπτυξης της στρατηγικής 2020 να έχουν ως ε, γνώμονα τον, τους νέους ανθρώπους. Η συμμετοχή των νέων σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες αλλά και στα πολιτικά πράγματα, είτε αυτό είναι σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, συμμετοχή των νέων στη θελοντική εργασία μέσω εθελοντικών οργανώσεων και επ' αυτού θα εκπονήσουμε και συμπέρασμα του Συμβουλίου συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών και στις άτυπες, ανεπίσημες μάλλον μορφές ε, δημοκρατίας. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα με καινοτόμο, διαφορετικό τρόπο. πολλοί νέοι άνθρωποι ε, δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε, στην εθελοντική εργασία και σε εναλλακτικές μορφές, αν θέλετε, δημοκρατικής συμμετοχή, συμμετοχή στα κοινά. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο έχουν μία διέξοδο να εκφράσουν την άποψή τους για τα τεκτενόμενα. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι νέοι αποκτούν μια σημαντική εμπειρία μέσω αυτών των εναλλακτικών μορφών ενασχόλησης με τα κοινά και με την εθελοντική εργασία. Το θεματολόγιο της Δανικής Προεδρίας για την νεολαία και την εκπαίδευση είναι αρκετά μακροσκελές. Αυτό θα απαιτήσει σημαντική δουλειά στο Συμβούλιο και ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν προκειμένου. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο εξάμεινο του 2012, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία στο Συμβούλιο και εμείς προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα εμεί και τη Προεδρία μα, ώστε να μπορέσει και η Κυπριακή Προεδρία να βασιστεί σε κάτι καλό. Σα ευχαριστώ και προσβλέπω στη συζήτηση μαζί σα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. διεξέλθει τα θέματα αυτά σε προηγούμενες συζητήσεις, ιδίως για τα θέματα της διαβίου ε, εκπαίδευσης που συνάπτεται με το αέρασμος για όλους. Ήταν μια σημαντική συζήτηση στην οποία εγώ επομίστηκα και την εκπόνηση της ε, αντίστοιχης ε, έκθεσης και έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και στην κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα. Η κυρία Εμπέρτ, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Υπουργό για την παρουσίαση της, ε, του προγράμματος, του φιλόδοξου προγράμματος της ε, Δανικής Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Θέλω να εκφράσω την ελπίδα ότι όλοι αυτοί οι στόχοι πράγματι θα μπορέσουν να επιτευχθούν μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Εγώ είμαι ευγνώμων σε εσά γιατί έχετε αναφερθεί στο θέμα του του έρασμου για όλους. Το όνομα αυτό δεν μας είχε αρέσει πάρα πολύ. Το θέμα βέβαια δεν είναι το όνομα, το θέμα είναι το περιεχόμενο. Και εγώ πιστεύω ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά <clears throat> για το καν κατά πόσο η έννοια αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση και αν κινδυνεύει να δημιουργήσει φρούδες προστοκίες στην κοινωνία μας. Επίσης είπατε ότι δεν είναι απαραίτητο να στεκόμαστε μόνο στην τυπική εκπαίδευση, θα πρέπει να σκεφτούμε και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης και δεν πρέπει να θεωρείται η εκπαίδευση μόνο σαν ένα, ένας προθάλαμος για την ε, εργασία, αλλά έχει, είναι αφ, αφεαυτού αξία, είναι πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ανάπτυξη η παιδεία. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με την κλασική ανθρωπιστική παιδεία είναι πολύ σημαντικά και σε ένα <clears throat> οργανισμό και, σε, και στον χώρο Εργασίες γιατί βοηθούν την πραγματική κατάρτιση και εξέλιξη ενός ανθρώπου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος Έρασμος για όλοι. <clears throat> Σίγουρα για τη δική μου πολιτική ομάδα αυτό είναι μια ιδιαίτερη μας διεκδίκηση ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα κομμάτι το οποίο να είναι σαφές και αναγνωρίσιμο ως ε, τμήμα της ε, εκπαίδευσης που δεν είναι μονάχα η τυπική εκπαίδευση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε και στις περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ μας. Η κυρία Τρουιπελ. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την ε, ομιλία σας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπατε για τη σημασία της παιδείας και του προπολογισμού για την παιδεία. Και είχατε ένα πολιτικό μήνυμα, να πούμε δηλαδή ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Και αν κατάλαβα καλά, αφήνεται όλο το ζήτημα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και του προπολογισμού στους υπουργού οικονομικών. Αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα κατά τη γνώμη μου. Εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε ή και μάλλον να ξεκαθαρίσουμε στους υπουργού οικονομικών ότι αν θέλουμε πραγματικά να, επιτύχουμε στη στρατηγική το 2020 και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της Ευρώπης και την ευημερία ε, των νέων, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στους υπουργού οικονομικών και πρέπει να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα σας προτείνω λοιπόν να ακολουθήσετε μία θαραλέα και επιθετική στάση. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, για τις ε, προτεραιότητες που έχετε αναφέρει σε σχέση με τη Δανική Προεδρία και θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο ελέγχθη προηγουμένως, το πόσο σημαντικό είναι για μας το πρόγραμμα Έρασμος και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια σύγχυση μεταξύ του πραγματικού του τωρινού προγράμματος Εράσμος και αυτού που θέλει να κάνει η Κομισιόν στο μέλλον. Για μένα το πρόγραμμα Έρασμος έχει πράξει πάρα πολλά υπέρ της ε, εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε συνθήκη. Το γεγονός ότι οι νέοι μας είχαν τη δυνατότητα να <clears throat> έχουν μια στενότερη επαφή χάρη στο πρόγραμμα αυτό, είναι κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό σύμβολο της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χαθεί αυτή η εικόνα. Είναι φυσικά σημαντικό και το θέμα της διαβίου εκπαίδευσης και αυτό δεν θα πρέπει να διαχυθεί σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, δεν ξέρω αν είναι στη δική σα αρμοδιότητα, είναι το θέμα τη επαγγελματική κατάρτιση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλιστεί απασχόληση για του νέου μα. Νομίζω σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη η επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι, ε, δεν έχει λάβει την έμφαση που θα έπρεπε και δεν της δίδεται η απαραίτητη αξία και ίσως θα πρέπει να κάνετε και εσείς μια προσπάθεια να δώσετε μια μεγαλύτερη ε, ορατότητα σε αυτή τη μορφή εκπαίδευση γιατί είναι σημαντική για τις θέσεις εργασίας. Κύριε Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφόσον έχουμε δανική, δανέζα, μάλλον υπουργό θα συνεχίσω στα δανεικά. Λοιπόν, Έχω μερικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ακούσατε ότι μας ανησυχεί το ζήτημα της ονομασίας. Ε, στους φιλελευθέρους εμάς δεν μας απασχολεί τόσο πολύ. Ε, κατανοούμε και οι πολίτε μα τα ξέρουν ε, περί τίνο πρόκειται. Εμείς πρέπει να ε, επιλύσουμε το κύριο ζήτημα του περιεχομένου και νομίζω ότι θα καταλήξουμε ένα συμβιβασμό. Αλλά το Εράσμου είναι το καλύτερο μπραντ εντό εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Συμφωνώ όμως με τον συνάδελφο Τουίβιλ για τον ε, ρόλο των Υπουργών Οικονομικών και το δικό μας ρόλο. Αν αφήνουμε όλα τα δημοσιονομικά ζητήματα στους Υπουργούς Οικονομικών, δεν παίρνουμε ούτε ευρώ. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Αλλά Εφόσον εδώ βρισκόμαστε στην Επιτροπή Πολιτισμού, θεωρώ ότι τα προγράμματα κινητικότητας, και αυτός είναι και μεγάλος στόχος για την Επιτροπή, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Μιλήσατε για μια εξέβρεση ισορροπίας και αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας στην ε, Δανέζικη Προεδρία. 73% αύξηση προτείνει η Επιτροπή. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Πού πιστεύετε θα καταλήξουμε. Χρειαζόμαστε μέσα, όχι μόνο ισορροπία, και μετά τα benchmarks που είπατε για την ε, απασχολησιμότητα. Είπατε ότι είναι δύσκολος αυτός ο τομέας. Μπορείτε αυτό να το αναπτύξετε λίγο παραπάνω. Θα θέλαμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά λοιπόν. Σας έχουμε καλή επιτυχία. Κυρία Πεναράπ. Ευχαριστώ για όλες τις ε, πληροφορίες, κυρία Υπουργέ. Έχω ορισμένα ζητήματα. Στα έγγραφό σας μιλάτε για τη στρατηγική για τι νέε δεξιότητε και τι θέσει εργασία, και είπε ότι θα μιλάμε για την επιχειρηματικότητα στην ε, κατάρτιση. Θεωρείτε ότι όλε οι καταρτήσει αυτέ θα επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες να γίνουν επιχειρηματίε, Δεν είναι ε, λίγο υπερβολικό αυτό. Ε, η κατάρτιση θα πρέπει να είναι πολύ πιο ευρεία. Υπάρχει βέβαια για το ζήτημα τη επιχειρηματικότητα, αλλά μπορούμε όλοι να γίνουμε επιχειρηματίε στο μέλλον. Μετά για την νεολαία, μιλάτε, λέτε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το πνεύμα δημιουργία και καινοτομία ε, για να προωθήσουμε την ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Αυτό είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά το ένα μεγαλύτερο ζήτημα και πρόβλημα είναι ε, η ανεργία στους νέους. Υπάρχουν νέοι που δεν ξέρουν, δεν έχουν που να μείνουν, ε, δεν μπορούν να διασφαλίζουν το μέλλον τους. Ποιες είναι λοιπόν οι συγκεκριμένες λύσεις που προτείνεται για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα της αβεβαιότητας στους νέους. Μετά για τη σύμβαση της UNESCO και την κύρωσή της. Τη στηρίζω απόλυτα αυτή την πρόταση. Πολλά μέλη δεν την έχουν ακόμα κυρώσει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύμβαση. Ε, αναφέρεται σε αυτή την ε, πολιτιστική ποικιλομορφία. Ε, η πρόεδρος λέει εδώ πέρα μιλάμε μόνο για την ε, εκπαίδευση, όχι για τον πολιτισμό. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. Ίσως μπορούμε να κάνουμε μια διακοπή να μπορέσει να απαντήσει η κυρία Υπουργός και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα που θέσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καμερβέρ για τις ε, ιδέες σας. Μιλήσατε για την αξία των άτυπων δεξιοτήτων. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό αν μπορούμε να συνδέσουμε, θα ήταν πολύ καλό αν μπορούμε να συνδέσουμε την ε, κατάρτιση, την διαβίου μάθηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πιστοποιήσει κάποιος τις δεξιότητες του για την αγορά εργασίας ε, και σας ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες σας. Ε, εντάξει, είναι λίγο σκληρός αυτός ο όρος ανθρώπινη πόρη, αλλά περί αυτού πρόκειται. Και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να αναφερθούμε στην εκπαίδευση και στην ανατροφή των ανθρώπων. Μιλήσατε για το Erasmus for All, αυτό το πρόγραμμα Erasmus για όλους. Θα επανέλθω και σε αυτό. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ όμως, σημαντικό και για το καθήκον που έχουμε αναλάβει, είναι να μην αφήσουμε την ονομασία ε, να έχει τον κύριο ρόλο εδώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια ιδιαίτερα φιλόδοξη λύση. Δηλαδή θέλουμε η εκπαίδευση να είναι το στοιχείο που θα μας οδηγήσει έξω από την κρίση. Παρατηρήσαμε ότι η ονομασία δίνει και ένα μήνυμα. Γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν είναι μόνο για τους ε, φοιτητέ. Πολλοί φορεί ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα. Εμείς ελπίζουμε ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια κατάλληλη λύση για το περιεχόμενο του προγράμματος. Πώς μπορούμε δηλαδή να επενδύσουμε στην γενετικότητα, στην ε, παιδεία, προς όφελος όλων των μορφών εκπαίδευσης και για τους νέους και για τους ενήλικες. Κυρία Τρίπλ. Με ρωτήσετε κάτι για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Είναι κοινό μυστικό βέβαια ότι η Ευρώπη, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια πολύ δύσκολη συζήτηση και οι συνάδελφοι υπουργοί και, και τα μέλη του Κοινοβουλίου και εδώ και αλλού θα εξακολουθήσουν να το συζητούν αυτό το ζήτημα στο επόμενο έτος. Το είπαμε και προηγουμένως ότι η κατάρτιση είναι ένας από τους κατάλληλους τρόπους να δώσουμε μια προοπτική για το μέλλον στους νέους αλλά είναι σημαντικό και οι νέοι να είναι προετοιμασμένοι για την είσοδό τους ε, στην αγορά εργασίας. Κατανοώ ότι θέλετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και μάλιστα μια δέσμευση σχετικά με, τους, με την επένδυση στον προπολογισμό. Αυτό θα το εξετάσουν οι υπουργοί στο ΕΚΟΦΗΝ. Δεν μπορούμε δηλαδή μόνο εμείς να το επιλύσουμε το ζήτημα. Υπάρχει βεβαίως υψηλό επίπεδο φιλοδοξία. Εμεί θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να υπάρξει πολιτική βούληση για την ε, εφαρμογή και του προγράμματος πλαίσιο. Αυτό πάντα όμως συνεργασία με τους συναδέλφους από το ΕΚΟΦΗΝ. Τώρα, για τον συνάδελφο Φίσας, αν προφέρω σωστά το όνομά σας, σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας για το Εράσμους και αυτή την ε, προοπτική της διαβιομάθησης. Σημαντικό στοιχείο αυτό και για μας. Και είπατε ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε συνολικά. Μία από τις λύσεις βεβαίως είναι εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση για τους νέους, αλλά υπάρχουν και ενήλικες που δεν έχουν αρκετές ε, δεξιότητες για να βρουν μια θέση εργασίας. Και αυτή είναι μια σημαντική πτυχή της ε, εκπαίδευσης. Η κατάρτιση των ενηλίκων, λοιπόν, δεν θα πρέπει να εξαφανιστεί ε, και να χάσει τη σημασία του αυτό το στοιχείο στο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Μιλήσατε και για την επαγγελματική κατάρτιση. Πολλές φορές μιλάμε για τις σπουδές των νέων, αλλά υπάρχει και επαγγελματική κατάρτιση και η σύνδεση της ε, εκπαίδευσης και της πρακτικής κατάρτισης, γιατί αυτό δίνει περαιτέρω δεξιότητες για το μέλλον και αυτό θα το εξετάσουμε κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης στις 24 και 25 Απριλίου στην Κοπενχάγη. Και εκεί ακριβώς ε, θα εστιαστούμε στην ε, επαγγελματική κατάρτιση μετά το σχολείο. Γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο μετά. Άλλη παρατήρηση Επίση για την ονομασία προγράμματος για ε, πρόγραμμα Εράσμου για όλους. Προφανώς αυτό απασχολεί πολύ κόσμο. Είναι σημαντικό, αναφέρθηκε, να μην μείνουμε μόνο σε αυτή τη συζήτηση για το πρόγραμμα. Όχι, πρέπει να συζητήσουμε από το περιεχομένο, αλλά είναι σημαντικό στοιχείο και η ονομασία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ιδιαίτερα τα κύρια στοιχεία, δηλαδή την επένδυση στην παιδεία. Αναφέρθηκα ήδη στα ζητήματα του προπολογισμού. το αναφέρετε κι εσείς, αλλά δεν αποτελεί τμήμα ε, ε, του δικού μας προγράμματος. Αυτό αποτελεί τμήμα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό και την οικονομία. Και τέλος, για την κυρία Μπεχνάχ. Μιλήσατε για την ε, καινοτομία και τη δημιουργία στην παιδεία. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι εμείς το έχουμε αναφε... Ε, συμπεριλάβει αυτό στο πρόγραμμά μας, στη Δανική Προεδρία. Θέλουμε αυτό να μας οδηγήσει ε, σε μια περισυλλογή για το περιεχόμενο της παιδείας. Και οι ίδιοι φοιτητέ, πέρα από την εκπαίδευση τους και την κατάρτισή τους, να αρχίσουν να σκέφτονται ε, να τους απασχολεί δηλαδή το ζήτημα της ε, κατάρτισης της και του περχομένου της. Μπορεί αυτό να γίνει βέβαια και μέσω μιας επιχείρησης. Ή στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Τώρα, ξέχασα ένα ερώτημα για τα benchmarks και την ε, επιλεξιμότητα στην αγορά εργασίας. Ελπίζω να απάντησα τα υπόλοιπα. Κύριε Λοκεγκάρτ, είπατε... Με ρωτήσατε μάλλον ποιοι είναι οι στόχοι της Δανικής Προεδρίας για την ε, ανάπτυξη τέτοιων ε, benchmarks. Δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί υπάρχουν ε, διαφορετικές μέθοδοι εργασίας των κρατών μελών. Εμείς θα θέλαμε να καθορίσουμε παραμέτρους για να δούμε πώς μπορούν οι νέοι να προετοιμάζονται καλύτερα για την αγορά εργασίας. Υπάρχουν βέβαια και διαφορές, αλλά είναι σημαντικό να δούμε πώς θα φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το σύστημα με τα benchmarks για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο. Και το ίδιο το μήνυμα είναι σημαντικό ότι θέλουμε να βρούμε τέτοια benchmarks. Αυτό είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που έχουμε να στείλουμε, ότι η κρίση είναι πολύ βαθιά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μέσα για να βρούμε την έξοδο και την προοπτική στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω άλλους πέντε Παρακαλώ, καλύψτε τα θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα καλυφθεί. Ο κύριος Μπάγκο. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, κυρία Μπενερά. Συνεχίζουμε τώρα. Ήταν ένα ερώτημα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Το θέμα της επισφαλούς θέσης στο οποίο βρισκόνται οι νέοι. Δεν απάντησε η κυρία Υπουργό στο θέμα αυτό. Øh, øh. ναι. Συγγνώμη που δεν απάντησα συγκεκριμένα στο ερώτημά σα. Νόμιζα ότι το είχα απαντήσει μαζί με τα ζητήματα καινοτομία. Ναι, πράγματι, είναι τρομερό το πώς οι νέοι αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι, δυσκολεύονται να βρουν μια θέση εργασίας, ε, ε, μεταναστεύουν για να έχουν καλύτερες προοπτικές στη θέση εργασίας. Εμείς θεωρούμε ότι το κλειδί εξακολουθεί να βρίσκεται ε, στην παλιά συνταγή, δηλαδή εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και μέσω των άτυπων μορφών εκπαίδευσης. Δηλαδή να βελτιώσουμε με διάφορους τρόπους ε, τις ε, δεξιότητες ε, των νέων. Βλέπουμε ότι πολλές φορές η κατάρτιση κάνει τη διαφορά. Πολλοί νέοι δεν έχουν μια θέση εργασίας, περιθωριοποιούνται και βλέπουμε και παρατηρούμε ότι αυτοί οι νέοι, ανεξαρτήτως από τις χώρες προέλευσή τους, έχουν χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν ήθελα να κάνω μια παρομοίωση θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν μια σχέση μεταξύ ατόμων που δεν έχουν ακριβώ την ίδια ηλικία. Ε, πάση τέθηκε το ερώτημα και απάντησε η κυρία Υπουργό. Εγώ θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ε, εξέβεσης μιας λύσης για να προωθήσουμε την εκπαίδευση, των, ε, την εκπαίδευση διαβίου μέχρι το 2014. Για το όνομα και για το περιεχόμενο του Εράσμου για όλους νομίζω ότι έχετε απαντήσει. Επομένως το μόνο θέμα το οποίο θέλω να ζητήσω και πάλι να διευκρινίσετε είναι η χρηματοδότηση των 17 εκατομμυρίων. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Και κάτι ακόμα, ο αθλητισμός. Υπάρχει ένα κεφάλαιο χωριστό για τον έρασμο στο, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Δεν έχετε όμως ε, δώσετε την ίδια, δεν έχετε δώσει την ίδια αυτονομία στον τομέα της νεολαίας. Κυρία Υπουργέ, έχετε παρουσιάσει φιλόδοξους στόχους, αλλά φιλόδοξοι στόχοι θέλουν και φιλόδοξη χρηματοδότηση. Το νέο πρόγραμμα Εράσμος για όλους <clears throat> βασίζεται στο ότι θα έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο των πολιετές από ό,τι στο παρελθόν. Και μόνο τότε έχει νόημα κάτι τέτοιο. Έχουμε προγράμματα για τη διαβίου εκπαίδευση, έχουμε προγράμματα για τον ε, έρασμο, έχουμε τονίσει τη σημασία της κινητικότητας μέσα στον έρασμο αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα και να τα συνενώσουμε αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες τομές να κινητοποιήσουμε και τους ε, ενδιαφέρομενους. Τι θα γίνει αν δεν έχουμε τη χρηματοδότηση. Έχει πράγματι νόημα το σχέδιο της Κομισιόν με τη μορφή που έχει τώρα ή θα ήταν καλύτερα να παραμείνουμε με τα προγράμματα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους και να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά τα οποία έχουμε για να συνεχίσουμε αυτά τα προγράμματα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο να υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτή η προσοχή δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα. Ένα δεύτερο σημείο, η επαγγελματική κατάρτιση αναφέρθηκε ήδη, απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε πάρα πολύ διαφορετικά συστήματα κατάρτισης και απόδοσης πιστοποιητικών για τα προσόντα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα μπορούσαμε να καταλάβουμε καλύτερα την θέση του καθενός, να έχουμε και μεταλαμβάνευση των πρακτικών. Θα υπάρξει μια συνδιάσκεψη για τα θέματα αυτά τον Απρίλιο, αλλά ακόμα ελείπει σε μεγάλο βαθμό η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχει η, το επίπεδο ε, εκπαίδευση στη Γερμανία που ονομάζεται Meister, το επίπεδο δηλαδή του τεχνίτη σε υψηλό επίπεδο που θα πρέπει αυτό ίσως να το ακολουθήσουν και άλλε ε, και άλλες χώρες. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρξει και ένα πνεύμα το οποίο θα υποστηρίξει αυτή την επαγγελματική κατάρτιση. Ο κύριος Μπόρης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Υπουργό που ανεφέρθηκε και στα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας για το γεγονός ότι συνεχίζεται και το έργο της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Η συνέχεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Θα θέλω να κάνω μια ερώτηση που αφορά την εφαρμογή όλων αυτών των πρωτοβουλειών. Ο έρασμο είναι σίγουρα ένα από το πλέον σημαντικό στοιχείο στην πολιτική σας και θα μας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη Προεδρίας σας. Θέλω να σα ρωτήσω για τις δικέ σας δεσμεύσεις του στόχου σας, γιατί πέρα από το Εράσμους τα κράτη-μέλη θα λάβουν ε, πολλά κονδύλια από τα διαφορετικά ταμεία που εν μέρη μπορούν να δοθούν στην εκπαίδευση και στην, στον εξυγχρονισμό της βάθμιας εκπαίδευσης και ουσιαστικά πρόκειται για κονδύλια που από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ρωτώ λοιπόν πώς θα μπορέσετε ή πώς προβλέπετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα χρήματα που μπορούν να δοθούν από τα διεθνωτικά ταμεία. Μια απάντηση γι' αυτό. Είναι αρμόδια για την εκπαίδευση, χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Μακλάκλιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Υπουργό για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις που δώσατε τώρα. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ναι, είναι η Επιτροπή Εκπροσωπή τους νέους. Είμαστε η φωνή των νέων για τις φιλοδοξίες και τους στόχους και θα θέλαμε να διαβάσουμε τις δικές τους ελπίδες σε εσάς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα το όνομα Έρασμος για όλους. Ε, το θέμα είναι να μειώσουμε την κρυφοκρατία και τα εμπόδια ε, που μάτια υπάρχουν και να αυξήσουμε την πρόσβαση ε, σε όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για του νέου και όπω είπε ο κύριο Φίσα που αναφέρθηκε στην επαγγελματική κατάρτιση, σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά την εμπειρία. Επίση, άλλοι συνάδελφοι μιλήσαν και για τι ανεπίσημε μορφέ εκπαίδευση. Θα θέλαμε, αν θέλετε ένα κάποιο ορισμό, τι είναι οι επίσημε, οι ανεπίσημε, οι άτυπε μορφέ εκπαίδευση, θα θέλαμε ε, να ορίσουμε καλύτερα αυτέ τι έννοιε. Θα ήθελα επίση να πω ότι μπορεί να μιλάμε για αρκετή ώρα για το τι θα ελπίζαμε και τις συμφιλοδοξίες μας ε, για τους νέους και τις δεξιότητές τους. Θα ήλπιζα πάντως η Ιδανική Προεδρία να επιλέξει ένα συγκεκριμένο στοιχείο, να θέσει ένα στόχο και να τον επιτύχει. Ποιο θα είναι το δικό σας benchmark ως Προεδρία. Και τέλος, για τον αθλητισμό. Υπάρχει ένας χωριστός προπολογισμό για τον αθλητισμό, ναι, ξέρουμε ότι είναι ειδινές οικονομικές στιγμές, αλλά επειδή ο αθλητισμός αφορά όλους τους ανθρώπους και όχι μία ελίτ μόνο, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες και πιστεύω ότι από αυτό το κονδύλι και τον αθλητισμό θα μπορούν να αποφεληθούν πολύ. Κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ πραγματικό λόγο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να πω για το εράσμος για όλους. Είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας. Και θα λέγα ότι τουλάχιστον θα πρέπει να αντιστρέψουμε τους όρους σε αυτήν ονομασία. Να πούμε όλοι για το εράσμος. Κατανοείτε τι λέω. Πρέπει βέβαια να εστιάσουμε πιο πολύ την προσοχή μας στο περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και όχι το σωστό όνομα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι Εσείς ως υπουργό για τα παιδιά και την εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό να σταθμίσουμε και να αξιολογήσουμε τις αξίες που έχουμε σε επίπεδο για αυτό το τομέα. Βεβαίως και τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά. Αλλά σε ό,τι αφορά τη στάση ζωή, τι συμπεριφορέ μα, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να περάσουμε κάποια καλά μηνύματα. Αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα είναι ο αποκλεισμό και οι διακρίσει. Βάσει τα στατιστικά στοιχεία, πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του αποκλεισμού, βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και πρέπει να βρούμε τρόπους να το εξαλείψουμε αυτό. Εξτρεμιστικά φαινόμενα, όπως αυτά που συνέβησαν στην Ορβηγία πέρυσι, είναι ανησυχητικά φαινόμενα. Μετά από τέτοια ε, τρομερά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, συζητούν ε, πλέον σε κάποιες χώρες μια πιο βασική νομοθεσία για την ε, οπλοκατοχή και οπλοκρισία. Αλλά χρειάζονται τέτοια τραγικά γεγονότα για να φτάσουμε εκεί. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τους νέους που επηρεάζονται α, ήδη από τα τρυφερά στάδια της ηλικία τους, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο τι νομοθετούμε και πώς εφαρμόζουμε την νομοθεσία και πώς χαράζουμε ειδικά την πολιτική παιδείας, γιατί επηρεάζουμε τον άνθρωπο, όπως είπα, από τα πρώτα στάδια της ζωής του. Δεν πιστεύω ότι να εστιάσουμε τόσο πολύ ή μάλλον μόνο στις δεξιότητες και στα προσόντα, αλλά σε κάτι γενικότερο, ώστε να μπορούμε να αποτρέψουμε τον αποκλεισμό. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρατήρηση ακόμα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε μαζί μου αν το θέμα των νέων και του αθλητισμού θα πρέπει να εξαιρεθεί από αυτό το πλαίσιο της διαβίω εκπαίδευσης. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει ιδιαίτερα με το γενικό πλαίσιο. Θα ήταν χρήσιμο να είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα. Η νεότης, ο αθλητισμός, να είναι ένα κοινό ένα κοινό σύμπλεγμα και θα ήθελα να έχω και την άποψή σας για το θέμα αυτό. Φυσικά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα στην Επιτροπή μας για όλα αυτά. Επίσης θέλω να σας παρακαλέσω να μας ε, συγχώρησετε βέβαια η κυρία Βασιλείου είχε τότε μιλήσει για το θέμα του να γίνει πιο ορατή η μη τυπική εκπαίδευση. Εγώ είχα μιλήσει τότε για το λεγόμενο ευρωδιαβατήριο το οποίο αφορά τα στοιχεία της μη αυτής τυπικής ε, εκπαίδευσης και εγώ είχα προτείνει να πάρει αυτό το όνομα του Ευρωδιαβατηρίου και η Ιρία Βασιλείου αναφέρθηκε σε ένα διαβατήριο για τους νέους. Τώρα να μην μπλεχτούμε με τα διαβατήρια, ναι, διαβατήριο νέων ή ναι, διαβατήριο δεξιοτήτων κτλ. Αλλά υπάρχει αυτός ο θεσμός και μπορεί να προσαρμοστεί στο να λάβει και άλλες μορφές γνώσεων όπως είναι η μη τυπική γνώση. Και θα ήταν χρήσιμο αν και εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για την επίτευξη αυτού του στόχου για την επαγγελματική κατάρτιση. Έχουν ελεγχθεί βέβαια πολλά, όχι μόνο στη Γερμανία και στην Αυστρία. Υπάρχει αυτό το διτό σύστημα, όπως γνωρίζετε. Και έχω μιλήσει και με τους Ισπανούς συναδέλφους. Τον Απρίλιο θα έρθουν στο Βερολίνο για να δουν ακριβώς πώς λειτουργεί στην πράξη το σύστημα αυτό εκπαίδευσης και κατάρτισης. Γιατί στη Γερμανία είναι στα 40% η ανεργία των νέων. Κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Πρέπει να βρούμε τρόπους λοιπόν και επίσης και η Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να βρει τρόπους ώστε να υπάρχει μια καλύτερη μεταλαμπάδευση των βέλτιστων πρακτικών. Συζητάμε για τα θέματα αυτά επί δεκαετίες, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά είναι τώρα τραγική κατάσταση σε ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία που είναι 40% η ενεργεία των νέων, αλλού 28%, σε εμάς είναι μονάχα 8%. Δεν μπορούμε λοιπόν <clears throat> να θεωρήσουμε ότι αυτά έχουν να κάνουν μονάχα με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά για το γεγονός ότι στη Γερμανία έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προωθεί τους νέους όχι μονάχα στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι ακολουθούν τέτοια χειρονακτικά πολλές φορές επαγγέλματα τα οποία όμως είναι ιδιαίτερα πρόσφατα. Για την αύξηση της χρηματοδότησης. 73% αύξηση, εντάξει θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά πάνω σε ποια βάση θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Όλοι θα πρέπει να αγωνιστούμε για κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να το κάνει μονάχα η Προεδρία του <clears throat> Συμβουλίου και δυστυχώς δεν είναι θέμα μονάχα των Υπουργών Πολιτισμού. Θα πρέπει να πάμε στους Υπουργούς Οικονομικών και να τονίσουμε ότι η κρίση που περνάμε και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι θα πρέπει να σημάνει ότι να σταματήσουμε τους δεκάρικους κυριακάτικους λόγους για την παιδεία και να δώσουμε πράγματι <clears throat> χρήματα και να κάνουμε επενδύσεις για την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Και τώρα για τον έρασμο προφανώς. Ο έρασμος έχει μια συμβολική σημασία, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό ε, σύνθημα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το πρόγραμμα αλλά είναι γνωστό όχι σαν όνομα μονάχα, αλλά γιατί εξασφαλίζει την κινητικότητα των νέων. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον τομέα αυτό. Υπήρξαν προτάσεις της Κομισιόν να υπάρχουν και δυνατότητε χρηματοδότηση και δανειοδότηση των φοιτητών οι οποίοι θέλουν να κάνουν ανώτερε σπουδέ, να κάνουν πρακτική εξάσκηση. Αλλά έχουμε βρει μια σειρά από προγράμματα όπως το Comenius το οποίο υπάρχει ήδη από το 1994 και το οποίο έχει και αυτό μια ζήτηση. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όλα τα πράγματα καλύπτονται από το Erasmus. Το Comenius έχει μια ανεξαρτησία και παίζει και κάποιο ρόλο για την ε, εκπαίδευση των ε, πιο μεγάλων στην ηλικία. Λοιπόν, δεν πρέπει να εξαφανιστούν αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν ε, αξία και να τα θέσουμε όλα κάτω από την ίδια οροφή. Λοιπόν, αν οι, οι δεν αγωνιστούν για προγράμματα αυτού του είδους, θα είναι κρίμα. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε Νομίζω ότι η Δανία έχει δώσει ένα πολύ καλό παράδειγμα στα θέματα αυτά και ε, εάν εσείς παρετηθείτε από τον αγώνα αυτό, εγώ θα συνεχίσω να σας πιέσω, γιατί εγώ δεν παρετούμε. Πρέπει μαζί με τους Δανούς στο επόμενο εξάμεινο να καταφέρουμε, να καταφέρουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές από την Κομισιόν. Η Κομισιόν βέβαια θα πρέπει να δώσει την απαραίτητη πολιτική εμβέλεια στα θέματα αυτά για να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η καλή πολιτική, όχι μονάχα να προτείνεται αυτό που θέλουν οι πολιτικοί. Πρέπει να υπάρξουν πρόοδοι και να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και είναι ωραία η ιδέα της διαβίου ε, εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η έννοια νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Which minister? Έχετε το λόγο. Ναι, ναι, δεν έχετε απαντήσει ακόμα, βέβαια. Ε, σωστό, το ξέχασα. Ήταν να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, δεν έχετε απαντήσει ακόμα. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. και για αυτή την ε, ιδιαίτερα ενθουσιώδη παρέμβαση στο τέλο. Ελπίζω και εγώ να καταφέρω να απαντήσω με τον ίδιο ενθουσιασμό στα ερωτήματα που μου θέσατε. Κύριε Μπάγκο, Εσείς και πάλι αναφερθήκατε στην διαβίου μάθηση και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αυτή είναι η κόκκινη γραμμή ή η κλωστή που συνδέει όλες τις παρεμβάσεις εδώ, ε, όλα όσα αναφέρατε εδώ, διαβίου μάθηση και πώς θα τη συνδέσουμε μαζί με την καινοτομία και ε, πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά πρακτικά. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες που έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της Προεδρίας μας. Αυτός ο συνδυασμός διαφορετικών αξιών. Ο κύριος Μπάκο επίσης ε, έθεσε ένα ερώτημα για τον προπολογισμό και σε αυτό, με αυτό βέβαια συνδέεται και ερώτημα άλλου συναδέλφου του κύριου Βερχόιεν για, το, για τον προπολογισμό και πάλι. Η Επιτροπή έχει υποβάλει μια φιλόδοξη και σημαντική πρόταση σε σχέση με την ε, νεολαία και την κατάρτιση και εκεί αναφέρεται το ποσοστό του 70%. Αύξηση δηλαδή του με το 70%. Αυτό έχουμε σημειώσει όλοι. Και σημειώνουμε ότι και πάλι ότι η παιδεία είναι πολύ σημαντικός τομέας που θα μπορέσει να μας ε, οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Ξέρουμε ότι επικρατεί βαθιά κρίση στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε όλα αυτά μακροπρόθεσμα. Βεβαίω, όμως από τώρα, από την Δανική Προεδρία, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή έχει και αυτή αποστείλει ένα χειρομήνυμα δήλωσε ότι αν υπάρχουν περαιτέρω φιλοδοξίες ε, στο ε, τομέα της παιδεία, τότε θα πρέπει να βρούμε και του κατάλληλου πόρου. Όμως αυτό ίσως μπορούμε να το αφήσουμε στους ε, αρμόδιους υπουργού. Τώρα, για την κυρία Βερχόγεν και η κυρία Μακλάρκεν και δύο αναφέρθηκαν στην σκοπιμότητα συγκεκριμένης αναφοράς ε, και καθορισμού των άτυπων δεξιοτήτων. Θα το εξετάσουμε ως Δανική Προεδρία, γιατί πράγματι ε, υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε την ε, σημασία ε, των άτυπων δεξιοτήτων και στο πλαίσιο της διαβιομάθησης. Και αυτό συνδέεται και με τα όσα θέλει να κάνει η Δανική Προεδρία για τις πραγματικές δεξιότητες. Όλα αυτά μπορούν να εξοπληθούν στην ε, κατάρτιση των υλίκων, στην διαβή μάθηση και ούτω καθεξής. Μετά ο κύριος Μπόρης έθεσε ένα ερώτημα για τα κοινωνικά ταμεία και τον ρόλο της παιδείας. Εμείς ως Προεδρία Ήδη αρχίζουμε να εξετάζουμε την ε, ε, διασύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και των κοινωνικών προγραμμάτων. Ήδη το έχουμε λάβει υπόψη λοιπόν αυτό. Κυρία Μακλάρκεν, ρωτήσατε κάτι και για τον αθλητισμό. Ελπίζω να επαναλάβετε το, το ερώτημα αυτό στον συνάδελφο Υπουργό Πολιτισμού. Γιατί είναι σε θέση να σας απαντήσει καλύτερα. Κύριε Τάκουλα, θα επιστρέψει? Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να, μπορώ να απαντήσω έτσι κι Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερος που βλέπω εδώ ανθρώπους ε, που για πολλά χρόνια έχουν εργαστεί στον τομέα της ε, παιδείας και πραγματικά κατανοούν ε, αυτό το πεδίο. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε ε, σε, στα άτομα που έχουν τις λιγότερες δεξιότητες. Αυτό ανέφερε ο κ. Στάκουλα. Και φτάνω και πάλι στην ενθουσιώδη παρέμβαση της Προέδρου και τα όσα είπε για το πρόγραμμα Grundtvig. Εξαιρετική ιδέα και εξαιρετική πρόταση, γιατί το Grundtvig ακριβώς αυτό αναφέρεται στις βασικές ε, δεξιότητες ε, και αυτό έχει μεγάλη επιτυχία και στη Γερμανία και αλλού. Θα ήθελα λοιπόν με την ε, ιδιότητά μου να πω ότι το Grundfig αναφέρεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα για μας, στην, στον τρόπο ζωής και στην νεοτροπία που θα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή για το αν θα συμμετάσχουν ε, στην διαβίου ή όχι. Θεωρούμε ότι όλοι οι ενήλικες θα πρέπει να συμμετέχουν. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο για το περιεχόμενο του και να μην ξεχνάμε τι, τι περιλαμβανόταν σε όλα αυτά τα προγράμματα, Γκρούντφιχ, Λεωνάρντο Νταβίντσι, Κορνίλιους. πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε όλα αυτά τα, διάφορα προγράμματα. Και έτσι αποκτούμε αυτή την συνολική και γενική άποψη. Και ο κύριος Τάκουλα είπε δεν πρέπει να λέμε Εράσμους για όλους, αλλά όλοι για το Εράσμους. Όχι μόνο για την ονομασία, αλλά και για το περιεχόμενο. Και ελπίζω ότι πράγματι θα είμαστε πιο αυστηροί και θα λέμε ξεκάθαρα πώς ε, θα διευρύνουμε τις προσπάθειές μας ε, για την παιδεία. Όχι δηλαδή μόνο με την ονομασία, αλλά και με το περιεχόμενο. Υπάρχουν βέβαια επιχειρήματα και για τις άλλες ε, μορφές και κατευθύνσεις της εκπαίδευσης, αλλά το περιεχόμενο είναι το πιο σημαντικό σε όλες αυτές τις ε, διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης. Το Φεβρουάριο θα ακόμα και μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα, για τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας σύνδεση της κατάρτισης με τις επιχειρήσεις και την, ε, τον περιορισμό της ενεργείας των νέων. Ευχαριστώ. Okay. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ε, τονίζω και πάλι το πρόγραμμα Grundfig θα πρέπει να τύχει μεγάλης προσοχής, σας το επιθυμίζω. Χαίρομαι για το γεγονός ότι ήταν τόσο ζωντανή αυτή η συζήτηση και βλέπω τα γελαστά πρόσωπα των συνεργατών σας που είναι πραγματικοί δανείοι, όλοι τους. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε ότι και τον επόμενο μήνα, τους επόμενους μήνες θα μπορούμε να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα επιτυχές πρόγραμμα για την ε, ε, διαβίου μάθηση. Ελπίζω ότι η Κομισιόν έχει αποκομίσει κάποιες ιδέες και γνώσεις και σας ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε για τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού από την Δανική Προεδρία και μου είπε η γραμματεία τόσο ωραίες είναι οι γραβάτες στους άντρες και ξαφνικά έρχονται άνθρωποι χωρίς γραβάτα εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό είναι αστείο τώρα, εσωτερικό αστείο της γραμματείας, απλώς σας το μεταφέρω, δεν νομίζω το είπε, για να είναι αγενής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας παρουσιάσω, μπορείτε να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας αμέσως. Ε, ναι, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, να πω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της κουλτούρας του καθενός και του πολιτισμού, αν θέλετε. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλούμε για πολιτισμό, δεν το παίρνω στραβά, είμαστε μέσα στο θέμα. Χαίρομαι ειλικρινά που ξεκινούμε με αυτό το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσωπικά το λέω, αλλά και ως εκπρόσωπος της Δανικής Προεδρίας για θέματα πολιτισμού. Θα ήθελα να πω ότι γενικότερα η πολιτική μας ε, και οι στόχοι που έχουμε θέσει απαιτούν ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτή. Στην ομιλία μου θα μιλήσω για τη δημιουργία της Ευρώπης, για τους Ευρωπαίους πολίτες, θα αναφερθώ στους εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς, τη φαρμακοδιέγερση, το τα στημένα παιχνίδια, τον εθελοντισμό στον αθλητισμό, πολλά λοιπόν είναι τα θέματα στον κατάλογό μου και περιμένω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια μετά. Είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι σήμερα μαζί σας. Ε, είχα επισκεφτεί βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα και είχα αρκετέ επαφέ με διαφορά μέλη, αλλά ω εκπρόσωπο του Συμβουλίου είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσλέπω πραγματικά συνεργασία μαζί σα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στενή αγαστή συνεργασία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίω μια τόσο δυσχερή οικονομική κατάσταση. Πρέπει να εξεύρουμε μια λύση, μια διέξοδο από την κρίση και πιστεύω ότι ο πολιτισμό θα μπορούσε να είναι μια τέτοια λύση. Ο πολιτισμός, οι τέχνες δημιουργούν μια συνεκτικότητα στην κοινωνία και ο αθλητισμό επίσης. Οι τέχνες, ο πολιτισμός, η δημιουργικότητα μπορεί να είναι η βάση για καινοτόμες λύσεις, νέους τρόπους σκέψης για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε καιρούς κρίσης. Οι νέες γενιές χρειάζονται ελπίδα για το μέλλον και ελπίζω ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα είναι τα κλειδιά για ένα καλύτερο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε όλοι όσο προς τώρα μπορούμε για να το κάνουμε αυτό πράξη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου και ιδίω η Επιτροπή Πολιτισμού. Λοιπόν, α σηκώσουμε τα μανίκια για να δούμε αυτές τις κοινέ προκλήσεις. Ο τίτλος, αν θέλετε, το σλόγγαν ε, της Δανικής Προεδρίας είναι ε, η Ευρώπη στη δουλειά. Ξεκινά τη δουλειά για να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να βγούμε από την κρίση. Βεβαίως, ε, πρώτη προτεραιότητα και μας είναι η συνεργασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες πρέπει να καταβάλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προγράμματα, της πρωτοβουλίας και τις προτάσεις μας Ξέρετε, υπάρχει και η σχετική πρόταση για την ε, δημιουργική Ευρώπη που ε, εμπεριέχει και την πρόταση και για τα οπτοκακουστικά μέσα. Λοιπόν, αυτή η πρόταση, η δημιουργική Ευρώπη, είναι κομβική σημασία για να δημιουργήσουμε ένα καλό πλαίσιο για την δημιουργία και τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Το Νοέμβρη ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε αυτή η πρόταση στο Συμβούλιο και η πρώτη συζήτηση έγινε το Δεκέμβρη. Η αρχική υποδοχή από τα κράτη-μέλη ήταν θετική. Βεβαίω υπάρχουν και επίμαχα σημεία, πάντω είναι υψηλή προτεραιότητα για την Προεδρία μα να ε, προωθήσουμε αυτή την πρόταση όσο γίνεται περισσότερο. Ο προϋπολογισμός βεβαίως εξαρτάται από τις γενικότερες διαπραγματεύσεις ε, που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ένωση για την περίοδο 2014-2020. Είναι ε, σίγουρο ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, αλλά στο Συμβούλιο του Μαΐου ελπίζουμε τουλάχιστον να υπάρξει συμφωνία του περιεχομένου πρόταση πρότασης και όχι ε, για τον προπολογισμό. Προσβλέπω συνεργασία και με το δικό σας ηγητή της Πολιτισμού και να πω ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα που θα μας απασχολήσει κατά το μας εξάμεινο που είναι η Ευρώπη και τους πολίτες. Σε τόσο ζωφερές οικονομικές ε, στιγμές, ε, ε, όπως αυτές που ζούμε, θα πρέπει να καταστήσουμε σημαντική την Ευρώπη για τους ε, πολίτες μας. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι κομμάτι της πραγματικότητας, της καθημερινότητάς τους η Ευρώπη. Ότι η Ευρώπη κάνει μια διαφορά. Και αυτό θα φανεί με την, τον τρόπο τον οποίο επενδύουμε και χρηματοδοτούμε πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την ε, προάσπιση και την προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό σε καιρούς κρίσης. Υπάρχει μία τάση, βεβαίως, σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς και κανείς να κλείνεται, αν θέλετε, στο καβούκι του και να χαρτίζεται από εσωστρέφεια. Γι' αυτό ε, μια από τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας μας είναι οι εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης στο Συμβούλιο θα συνεχίσουμε τις εργασίες ε, βασιζόμενοι στην εξαιρετική δουλειά που έκανε η Ουγγρική και η Πολωνική Προεδρία. Θα έχουμε πολλές επαφές με υψηλόβαθμους ε, εκπροσώπους σε θέματα πολιτισμού και εξωτερικών σχέσεων από τις ε, τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Θα έχουμε σχετικές εκδηλώσεις στην Κοπενχάγη την Άνοιξη για να μπορέσουμε να καθορίσουμε καλύτερο τρόπο του πολιτισμού στι εξωτερικέ μα σχέσει. Είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Σάκα και την ενδιαφέρουσα έκθεσή τη για το θέμα αυτό και ελπίζω το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην διάσκεψη τη Κοπενχάγη. Η γενικότερη διάδραση με τον έξω κόσμο γίνεται πιο εύκολη με τις εξελίξεις και την ανάπτυξη του, ε, της ψηφιακής τεχνολογίας. Έτσι έχουμε ε, πιο εύκολα προσπελάσιμα μουσεία, βιβλιοθήκες όλο τον κόσμο και διάφορες ε, συλλογές ε, είναι πιο κοντά στον πολίτη. Η ψηφιοποίηση λοιπόν της πολιτικής κληρονομιάς ε, δραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί επιτρέπει στον κάθε πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο χρειάζεται, ανα πάσα στιγμή. αν λοιπόν ψηφιοποίηση και η αποθήκευση και διαχείριση του πολιτιστικού υλικού ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε όλους ε, τους ενδιαφερόμενους από το πρόγραμμα Europeana ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και προτεραιότητα για μας. Σε... Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της ψηφιοποίησης της πολιτικής κληρονομιάς, εμείς είμαστε της γνώμης ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει την ε, σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά και αυτό θα το κάνουμε με μια δέσμη ε, συμπερασμάτων ε, του Συμβουλίου. Κάτι άλλο που μας απασχολεί ιδιαίτερα και προσβλέπουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός που πλέον συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη και άρα θα πρέπει να υλοποιήσουμε το πρώτο ευρωπαϊκό ε, σχέδιο δράσης για τον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο χρόνο. Και εδώ αναφέρουμε και σχετική έκθεση του κυρίου Φίσας για την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό. Το πρόγραμμα εργασίας μας ε, Υπάρχει ένα κεφάλαιο για την ακαιρεότητα στον αθλητισμό, κάτι πολύ σημαντικό που μας απασχολεί όλους. Όλοι γνωρίζουμε το φαινόμενο της φαρμακοδιέγερσης και το στήσιμο των παιχνιδιών, κάτι που καταφέρει κέριο πλήγμα ε, στον αθλητισμό, που συνήθως προσφέρει σημαντικά πρότυπα στην κοινωνία. Η καταπολέμηση λοιπόν του ντόπινγκ και των παράνομων στοιχημάτων και του στήματο του παιχνιδιών είναι κάτι πολύ σημαντικό για μα. Υπάρχει πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βεβαίω για τον Εράσμος για όλους και υπάρχει ένα κεφάλαιο για τον αθλητισμό είναι προκειμένου. Θεωρούμε λοιπόν το, το κεφάλαιο του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό σκέλος της πρόταση αυτή και είμαστε δεσμευμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ιδανική Προεδρία σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό ειδικά, θα προσπαθήσει να δει το θέμα όσο γίνεται πιο αμερόληπτα και θα προσπαθήσει να έχει τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των ενδιαφερομένων. ο εθελοντισμός και ο εθελοντισμός στον αθλητισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνιστόσα και είναι στοιχείο συνοχής ε, για οποιαδήποτε κοινωνία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προωθήσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Να σας πω ότι υπάρχει και πρωτοβουλία Sport Vision 2012 που θα εστιάσει στην εθελοντική έργα στον αθλητισμό, τη φαρμακοδιέγερση και τον αθλητισμό ε, για όλου. Είναι μια εκδήλωση που θα λάβει η χώρα στην Κοπεχάγη το Μάρτιο και ελπίζω να είσαστε και σε εκεί. Εμεί βεβαίω θα εστιάσουμε πιο πολύ στι εργασίε εδώ στι Βρυξέλλε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική στι διαπραγματεύσει για όλε τι ε, πρωτοβουλίε που ανέφερα ε, νωρίτερα. Και βεβαίω θα δώσουμε έμφαση και εσωτερική διάσταση του πολιτισμού και του αθλητισμού και περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα για την επίσημη επιλογή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2016. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τα θεμέλια, καλά θεμέλια, για την Κυπριακή Προεδρία που θα έρθει μετά από εμά. Δράτω τι ευκαιρία για να ευχαριστήσω ε, του Πολωνούς και κυπρίου συναδέλφου και την εξωτερική συνεργασία που είχαμε στη τρία των Προεδριών. Σα ευχαριστώ επίσης εσάς, όλους εσά, τα μέλη τη Επιτροπή Πολιτισμού και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη. Πιστεύω ότι είναι η ώρα για ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Η κυρία Τρίπελ τώρα θέτει το πρώτο ερώτημα. Ευχαριστώ Ντόρις, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία που θίξατε. Μιλήσατε για το ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές μας σχέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικός και προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή προσέγγιση, το σωστό ύφος, τη σωστή διατύπωση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας προσέγγιση για τις χώρες της Μεσογείου, τις αραβικές χώρες της Μεσογείου και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη δημοκρατική πορεία στις χώρες αυτές, γιατί φυσικά αυτό είναι ένα κομβικό θέμα αυτή τη στιγμή, να μην σταματήσουμε την υποστήριξή τους. Θέλω λοιπόν να ξέρω τι θα κάνει η Ιδανική Προεδρία σε σχέση με το θέμα αυτό. Μίλησατε στη συνέχεια για την ψηφιοποίηση του καλλιτεχνικού των καλλιτεχνικών προϊόντων, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε αρχεία καλλιτεχνικών προϊόντων. αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε να, βρούμε, να αντιμετωπίσουμε νέους τρόπους να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του copyright για τα θέματα αυτά. Έχει κλείσει η πρόσφατα με δικαστική απόφαση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας προσέγγιση ως Δανικής Προεδρίας. Ο κύριος Μπόρις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση αυτή και για το γεγονός ότι έχετε ε, αποφασίσει να συνεχίσετε την εργασία της προηγουμένης Προεδρίας της ε, Πολωνίας. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατά πόσο το έγγραφο ΑΚΤΑΤ για τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών θα εξακολουθήσει να είναι μια έγκυρη πρόταση. Τι θα κάνει λοιπόν η Προεδρία της Δανίας, η Δανική Προεδρία για το θέμα αυτό ακτά. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι ένα από τα αντικείμενα της δικής σας Προεδρίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας ε, δείξω και φυσικά <clears throat> υποστηρίζω απόλυτα τη στάση σας είναι το θέμα των προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο να τονώσουν την δημιουργικότητα στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα «Η Δημιουργική Ευρώπη» παραδείγματος είναι απαραίτητο να έχει μια αυτονομία το κάθε ένα από τα συστατικά του στοιχεία, αυτό που αφορά τα μέσα ενημέρωσης και αυτό που αφορά τον πολιτισμό. Νομίζετε λοιπόν ότι θα δώσετε μια μεγαλύτερη αυτονομία σε αυτά τα δύο υποπρογράμματα που βρίσκονται στα πλαίσια της Δημιουργικής Ευρώπης και κάτι ακόμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν συζητήσετε με τους υπουργού <clears throat> πολιτισμού και θέλετε να αποφασίσετε για το περιεχόμενο των προγραμμάτων πολιτισμού θα τεθεί και το θέμα των ε, διαθωτικών πόρων, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ που μπορούν να κατευθυνθούν προς την υποστήριξη του πολιτισμού από τα διαρθρωτικά ταμεία και αυτό μπορεί να βοηθήσει και τις περιφέρειες της Ευρώπης να προωθήσουν τα πολιτιστικά θέματα. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής διαρθρωτικού χαρακτήρα θα αγωνιστείτε για να έχει και ο πολιτισμός ένα ρόλο στα διαρθρωτικά αυτά ταμεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Κύριος Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Υπουργό. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα ενημασίας, εγώ θα εκφράσω αλληλεγγύη προς το πρόσωπό σας. Και καταγράφω τα σχόλια της Προεδρίας, αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν φορά ή όχι γραβάτα αλλά τι γραβάτα φορά. Ξέρετε, η Ιδανική τι γραβατα φορα έχει μοιράσει μια εξαιρετική γραβάτα ως δώρο, αλλά εγώ τη βρίσκω κάπως βαρετή παρά τα αυτά. Λοιπόν, κάποια σχόλια και μια ερώτηση προ τον Υπουργό. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία Ευρώπη για τους πολίτε θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Δεν γνωρίζω όμως κατά πόσον Κύριε Υπουργέ, έχετε, έχετε σημειώσει το, το Κοινοβούλιο δεν ε, προβλέπεται να μπει στη διαδικασία απόφαση, οπότε δεν έχει λόγο εν προκειμένου. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι αρκετά λυπηρό. Η νομική βάση της, ε, που, επι, που επελέγει στο Συμβούλιο είναι το άρθρο 256. Κατ' εμέ είναι ακατανόητο αυτό. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για τους πολίτες, ε, πώς δεν έχει λόγο ε, και μέρος, αν θέλετε, σε αυτή την ε, απόφαση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν το κατανοώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει κοινωνός της διαδικασίας λήψης απόφασης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για αυτό το φάκελο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο πολιτισμός, ευρωπαϊκός πολιτισμός και η σχέση με τον ε, λοιπό κόσμο. Πολλοί συνάδελφοι και κυρία Τρίπο αναφέρθηκαν στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, που βεβαίως είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και είναι θέμα επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θα αναφερθώ στην Κίνα και τις σχέσεις της Ένωσης με την Κίνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις αυτές. Σε μια χρονική συγκυρία προσπαθούμε να δώσουμε όθεση στην ανάπτυξη, αλλά και να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις μας με την Κίνα. Η Κίνα αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τρίτο πυλώνα στις εξωτερικές της σχέσεις και αυτός ο τρίτος πυλώνας αφορά την πολιτιστική συνεργασία. Υπάρχει λοιπόν ο πρώτο πυλώνα που αφορά την πολιτική, ο δεύτερο την οικονομία και ο τρίτο ο πολιτισμό. Γιατί λοιπόν ε, να μην ε, εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να έχουμε μια πολιτιστική συνεργασία και με την Κίνα. Μπορεί να έχουμε και εμείς κάποιο ωφέλη από αυτό. Πιστεύω ότι η Επιτροπή και η κυρία Βασιλείου που έχει επισκεφτεί την ε, Κίνα αρκετές φορές, αλλά και εμείς η Επιτροπή Πολιτισμού, μπορούμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας απευθύνω μια έκκληση εν προκειμένου. Και επιτρέψτε μου και μια, ένα μικρό παράπονο ε, για τα θέματα επικοινωνία, καθώς είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπής μας και η επικοινωνία. Η Προεδρία σας, εσείς κύριε Υπουργέ, θα θέσετε το θέμα της βελτίωσης επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι κομμάτι των προτεραιότητων σας Προεδρία. Και τέλος, για τον αθλητισμό. Τα στημένα παιχνίδια και η φαρμακοδιέγερση είναι πολύ σοβαρά θέματα συμφωνώ με το γεγονός ότι τα θέσετε ως προτεραιότητα. Όμως και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο και η όλη Ένωση, όλοι πιστεύω και η Προεδρία, θα ήθελα να εστιάσουμε και πολύ στον αθλητισμό και τη δημόσια υγεία, γιατί η δημόσια υγεία εξίσου είναι ένα θέμα. Και στη Δανία και αλλού ήδη τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, πώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει σημαντικά εντυπωσιακά στη βελτίωση της υγείας. Να, ένα τομέα, η δημόσια υγεία, όπου έχουμε πολύ υψηλές δημόσιες δαπάνες Και να, λοιπόν, μια ευκαιρία που μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι χρειάζονται πρωτοβουλίε σε αυτό το τομέα. Ρωτώ λοιπόν, η Προεδρία προτίθεται να κάνει κάτι για αυτά τα δύο. Κυρία Καμέρα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για τις παρατηρήσεις τους, του. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη διέρχεται μια κρίση, είναι όλο και πιο εντυπωσιακό και Ανησυχητικό βέβαια το, βλέπουμε, το να βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει όλο και λιγότερη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ελπίζουμε ότι με τον πολιτιστικό χώρο και ιδίως με τα νέα προγράμματα για τον αθλητισμό θα υπάρξει μια <clears throat> μεγάλη βοήθεια να μπορέσει να τονωθεί αυτή η ευρωπαϊκή κουλτούρα, γιατί αυτό είναι ο ελίπων κρίκος, σύμφωνα με την ε, άποψή μου. Είναι μια πολύ σημαντική λοιπόν πτυχή που πρέπει να την προωθήσουμε και στη δική μας ε, Επιτροπή φυσικά με τη βοήθειά σας. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μπόρις, αναφέρθηκε και στο Ταμείο Πολιτισμού. Ξέρουμε ότι για τον πολιτισμό και για τον αθλητισμό δεν πρόκειται μονάχα στο να υποστηρίξουμε συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια, αλλά πολλές φορές πρέπει να δημιουργήσουμε και τις απαραίτητες υποδομές. Και άμα δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι η κατάσταση με τους ε, δήμους, με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που θέλουν να υποστηρίξουν τέτοια σχέδια για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, ξέρουμε ότι τους λείπουν τα χρηματοδοτικά μέσα. Επομένως, θα ήταν απαραίτητο να εξασφαλίσετε μέσα και από τα περιφερειακά ταμεία να εξασφαλίσετε ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός θα παίζουν κάποιο ρόλο, ιδίω μέσα στα μέτρα δημιουργία <clears throat> υποδομών και να την χάνουν χρηματοδότηση, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και να την υποστηρίξουμε για να προωθήσει τα θέματα του προπολογισμού του πολιτισμού συγγνώμη, και του αθλητισμού και θα είναι σαφές ότι εδώ η Ευρώπη πράγματι παίζει ένα θετικό ρόλο για να υπάρξει μεγαλύτερη ενσωμάτωση και μεγαλύτερη συνεργασία μέσω του πολιτισμού και του αθλητισμού και όλα αυτά φυσικά θα συμβάλλουν στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας για τους πολίτες μας. Θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη και γι' αυτό σας ευχαριστώ για το, την πρόθεσή σας να υποστηρίξετε μια τέτοια πορεία. Ο κύριος Μπέλτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την ομιλία σας. Με κάθε σεβασμό και το ζήτημα της αγεραιότητας ε, που έχει κεντρικό ρόλο στην Δανική Προεδρία, αρχικά Μόρτεν πρέπει να πω ότι συμφωνώ μαζί σου για τη σύνδεση μεταξύ αθλητισμού και νεολαίας και με το σε την πτυχή ε, της έκθεσης εντεγωφής από αφορά τον αθλητισμό αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ακαιρεότητα και έχω ορισμένα ερωτήματα εδώ για σας κύριε Υπουργέ. Είπατε εδώ ότι αποτελεί προτεραιότητα για σας, αλλά πιο συγκεκριμένα για τους πράκτορες των παικτών υπήρξε μια εξαιρετική διάσκεψη πρόσφατα και τα πολύ ενισχυτικά στοιχεία και αποτελέσματα της μελέτης των ε, υπηρεσιών της Επιτροπής από δύο χρόνια για τους πράκτορες. Υπάρχει λοιπόν αρκετή αβεβαιότητα για την ε, για τους πράκτορες των αθλητών και υπάρχει ζήτημα και με την αγκαιρότητα γενικότερα του τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω αν εσεί ε, έχετε σκοπό να αναλάβετε αυτή την πρόκληση γιατί υπάρχει αυτορύθμιση στον ε, τομέα των διαφορεμένων μερών, αλλά όταν αυτό δεν είναι επαρκές, γιατί αυτό το βλέπουμε αρκετά χρόνια τώρα, αν είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε μια πρωτοβουλία, βεβαίως μαζί και με την Επιτροπή, για να ασκήσετε πιέσεις σε αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βεβαίως έχουν γίνει κάποιες αναφορές ε, ε, στην ε, καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης και των στιμένων παιχνιδιών. Βεβαίως πολύ σημαντικό. Περιμένουμε μια απόφαση μάλλον την επόμενη Δευτέρα. Είναι σημαντικό να διαλέξουμε στρατόπεδο και εδώ. Ξέρουμε την θέση της Βάντα και θα θέλαμε να μας πει η Δανική Προεδρία αν ε, θα τη στηρίξει και θα στηρίξει και την ε, χρήση όλων των κατάλληλων τεχνολογιών στην μάχη αυτή κατά της φαρμακοδιέγερσης. Συμφωνείτε με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει όλες αυτές τις διαθέσιμες τεχνολογίες, γιατί ε, και η φαρμακοδιάγηση και τα στημένα παιχνίδια απειλούν την ακαιρεότητα και την αξιοπιστία του αθλητισμού. Και θα θέλαμε να το θέσετε ως ε, πραγματική προτεραιότητα και πιο συγκεκριμένα. Ε, Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό για την τοποθέτησή του και ιδίω ε, γιατί έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης ε, το πόσο ο πολιτισμό μπορεί να συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση που ζούμε. Επισημένοντα πώς οι πολιτιστικοί θεσμοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν λιγότερες ε, συνέπειες από την ε, κρίση και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ε, καταγράψει και κάποια κέρδη. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής ε, που αφορά την Δανική Προεδρία και θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα και αναφέρομαι στον προπολογισμό. Και τρία επιμέρους ζητήματα. Πρώτον, η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα θέμα που πιστεύω μας απασχολεί όλους ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε σήμερα. Πόσες ανάγκες για παρεμβάσεις υπάρχουν, για προστασία και α, έργα βελτίωσης ε, για τα πολιτιστικά μας μνημεία χρειάζονται. Σε ό,τι αφορά τον φιλτισμό, ε, θα έλεγα ότι δεν θα είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι ο πολιτισμό θα πρέπει να είναι κομμάτι ε, τη ίδια πρωτοβουλία για θέματα πολιτισμού. Ε, σε, πάθε, σε κάθε περίπτωση, ρωτώ ποιε είναι οι επιμέρου συγκεκριμένε πρωτοβουλίε τη Δανική Προεδρία, εν προκειμένου. Και τέλο, για τον εθελοντισμό. Αναφερθήκατε στον εθελοντισμό, ναι. Το 2011 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτο ε, Εθελοντισμού και είναι ο εθελοντισμό ένα από τα ζητήματα που αγγίζει πολλού τομεί. Ρωτώ, πώς προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε, αυτή την ευκαιρία που σας δίνετε, καθώς οι νέοι ε, είναι πολύ εθελοντές. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την ευκαιρία που ε, είχαμε να ε, έχουμε κάποιες επαφές στα τέλη της προηγουμένης χρονιάς και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όχι γιατί για μένα ο πολιτισμό ε, δεν είναι σημαντικό, το αντίθετο, αλλά θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στον αθλητισμό και να θέσω κάποια ερωτήματα. Η έκθεσή μα υιοθετήθηκε με 28, 28 ψήφου υπέρ και 8 κατά και ελπίζουμε να υιοθετηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Ολομέλεια που θα λάβει η χώρα εδώ στι Βρυξέλλε. Ήδη πολλοί συνάδελφοι σχολίασαν τα θέματα αθλητισμού θα ήθελα και εγώ να επιμείνω σε κάποια ζητήματα που πιστεύω ότι απαιτούν νομοθετικές αλλαγές στα κράτη-μέλη της Ένεσης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που απαιτεί μια δυναμική που πρέπει να δώσει Προεδρία. Η διαφθορά στον αθλητισμό, το θέσατε. Τα στοιχήματα, πρώτα στοιχήματα, όχι μόνο όμω αυτά, αλλά και η διαφάνεια στα πλαίσια των αθλητικών Εθνικών Ομοσπονδιών, των Εθνικών Ομοσπονδιών, Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και η διαφθορά και η πάταξή της ε, απαιτεί διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ε, προϊόντων φαρμακοδιέγερσης αυτό λειτουργεί παράλληλα όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Δηλαδή για μέ το μείζον σε ό,τι αφορά το ντόπινγκ είναι το πώς μπορούν να επηρεάσουν τα γυμναστήρια, τα σχολεία και η αεραστεχνική αθλητική σύλλογη προκειμένου και πώς θα πρέπει να υπάρχουν ποινικέ κυρώσεις για την χρήση τέτοιων ουσιών. Θα πρέπει, πιστεύω, να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ένωσης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της βίας, της διακριτικής μεταχείρισης, την αντιμετώπιση των χούλιγκαν και των φανατικών οπαδών ε, των ομάδων, ώστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ε, ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και μπορεί να αποτελέσει και πηγή ε, ενσωμάτωσης και ένταξης πολλών κοινωνικών ομάδων. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά ταμεία, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ιδιωτικά ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον πολιτισμό αλλά και για τον αθλητισμό. Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια στη διαθεσή μα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα να πούν ρητά πώ θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια πολύ ε, πιο σαφώ από ό,τι σήμερα. Ε, ε, Κύριε Υπουργέ, το θέμα του πολιτισμού και η ψηφιακή ατζέντα είναι κάτι το οποίο αναφέρατε. Εν συντομία, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό το θέμα και να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφιακή ατζέντα δεν αφορά μονάχα την εξασφάλιση των πολιτιστικών αγαθών, αλλά είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άτομα που έχουν δημιουργικό χαρακτήρα και μπορούν να δείξουν το πόσο δυναμική είναι η πολιτιστική βιομηχανία στην Ευρώπη και να έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία τα προϊόντα τους. Πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζεται η ψηφιακή ατζέντα μονάχα με την οπτική γωνία της εμπαραγματοποίησης των τεχνικών πλευρών και δεν λαμβάνει υπόψη επαρκώς η πολιτιστική πτυχή. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα για την συζήτηση που θα πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια, το θέμα του copyright, το θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου, όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν επίσης με την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων, τα ε, μοντέλα τα οποία είναι ανεξάρτητα από την τερματική συσκευή, αν είναι smartphone ή αν είναι υπολογιστές, tablet κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα ανακύψουν στους επόμενους μήνες, πιστεύω, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι καυτά θέματα συζήτησης. Αυτά δεν συζητώνται πολλές φορές και υπό την πολιτιστική έποψη, γιατί τα πολιτιστικά αγαθά δεν είναι μονάχα τα υπάρχοντα αγαθά που πρέπει να προστατεύσουμε, αλλά και οι νέε μορφέ δημιουργικότητα που μπορούν να προκύψουν. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο μέσα στου στόχου τη Δανική Προεδρία είναι να ενσωματώσουν και το θέμα του πολιτισμού περισσότερο στην ψηφιακή αζέντα. Τέλος, κυρία Μπεναράπ, ατού. Euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Θα επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά μου λοιπόν. Στο έγγραφο που μας στείλατε αναφέρεται ότι η Προεδρία έχει θέσει ως στόχο να παρακολουθήσει την κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της UNESCO. Πολύ σωστή κίνηση, αλλά με ποιο τρόπο θεωρείτε με ποιο τρόπο σκοπεύετε να ε, προχωρήσετε. Συμφωνώ με τον κύριο Λόγκεγκαρτ. Θα ήθελα να ξέρω εάν θα εργαστείτε για την εφαρμογή της συναπόφασης ε, με το Κοινοβούλιο στον τομέα του πολιτισμού. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Και τώρα τέλος, για το πολιτιστικό τομέα ω τομέα δημιουργία θέσεων εργασία. Είπατε ότι θέλετε να βγούμε από την κρίση, ότι ο πολιτισμό είναι ένα, μέτρο, με ένα μέσο που μπορεί να μα βοηθήσει, πράγματι, αλλά είναι και τομέα όπου υφίστανται θέσει εργασία αυτή τη στιγμή, που θα μπορούμε να το στηρίξουμε. Και θα ήθελα να ξέρω αν έχετε θέσει τέτοιο στόχο, όπω και να έχει, εγώ σα παροτρύνω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχετε κάνει λάθος. Υπάρχει συναπόφαση στον πολιτισμό. Δεν υπάρχει συναπόφαση στον... Ε, στην ηθαγένεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν για τις ερωτήσεις. Ε, πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, ελπίζω να τις κατάλαβα καλά, θα με βοηθήσει και η Πρόεδρος. Αρχικά, το ερώτημα της κυρία ε, Τρίπον για τον πολιτισμό και τη... σε ό,τι φορά και τις τρίτες χώρες. Είναι και για μένα προσωπικά και για την Προεδρία πολύ σημαντικό στοιχείο. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πολιτιστική συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Ένα καλό παράδειγμα είναι και ε, η Αραβική Άνοιξη και τα όσα συμβαίνουν στην ε, Μέση Ανατολή. Πώς μπορούμε να ε, στηρίξουμε αυτό το δημοκρατικό κίνημα. Είμαι πεπισμένος και έχω και προσωπική εμπειρία μάλλον για το πώς μπορούμε να ε, ε, χειριστούμε τέτοιες ε, καταστάσεις και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τέτοια κινήματα τόσο σε αυτές τις χώρες όσο και αλλού στον κόσμο. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και για την πρόθεση του πολιτισμού να διαμορφώσουμε επαφές αν θέλετε με τον πολιτιστικό χώρο της ε, κάθε χώρας και μπορούν να έχουν την ίδια σημασία με τις επίσημες επαφές που υπάρχουν με αυτές τις χώρες. Για τον κύριο Λόκακορν, και εσείς ε, θέσατε ένα ερώτημα για την Μιλήσατε για τις σχέσεις μας με, με τους ε, γείτονές μας, τις αραβικές χώρες, αλλά και με τις ε, σχέσεις μας με την Κίνα. Πολύ σημαντικές οι σχέσεις αυτές, πράγματι. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να προσπαθούμε να δημιουργούμε ε, σταθερές επαφές. Εγώ πριν από δέκα μέρες μόλις ήμουν στο Πεκίνο και συνομίλησα με τον Υπουργό Πολιτισμού της Κίνας και ήδη προγραμματίσαμε μια συνάντηση εδώ στις Βρυξέλλες όπου θα πούμε ξεκάθαρο ότι η πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ευρώπης είναι πολύ σημαντική. Χθε ε, που έφτασα εδώ στο ξενοδοχείο είχα ήδη μια μεγάλη στίβα εγγράφων ε, και εφημερίδων της Κίνας, όπου υπήρχε αναφορά στην συνάντησή μου με τον, με τον Υπουργό Πολιτισμού εκεί. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις φιλοδοξίες ε, που θέτουμε για μια τέτοια συνεργασία. Και υπάρχουν διάφορες παράμετροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μιλάμε και για τα δημοκρατικά αυτά και για τον επιχειρηματικό κόσμο και για την επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει να δούμε πώς θα εξετάσουμε και την πολιτιστική πτυχή όλων αυτών. Βεβαίω και η Δανική Προεδρία έχει υψηλέ φιλοδοξίε σε αυτό το τομέα. Η κυρία Τρίφελ επίση αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση και στα πνευματικά δικαιώματα. Αρκετά μέλη τη Επιτροπής αναφέρθηκαν σε αυτό. Είναι βέβαια ευαίσθητο το ζήτημα. με δύο ζητήματα κυρία σημασία. Πρώτον, λέμε ότι πρέπει να είναι όλα τα στοιχεία δωρεάν και να δώσουμε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. Και με, από την άλλη, πρέπει να προστατεύσουμε και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και καλλιτεχνών. Η Προεδρία θεωρεί σημαντικό να τονίσουμε την κλοπή που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Ε, σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά αγαθά. Είτε πρόκειται για μουσική, για κινηματογράφο, για ηλεκτρονικά βιβλία. Εάν θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη μια ισχυρή πολιτιστική βιομηχανία, θα πρέπει να, να φροντίσουμε ε, να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των δημιουργών. Ιδάλλως δεν γίνεται να έχουμε μια ισχυρή βιομηχανία και αυτό τα κρίμα γιατί υπάρχει ε, δυναμική ανάπτυξη σε αυτές τις βιομηχανίες εδώ. Εμείς λοιπόν βρούμε προτεραιότητα αυτό το ζήτημα και ξέρουμε ότι διεξάγεται συζήτηση σε πολλές χώρες ε, στην εξέβρεση μιας ισορροπίας για ε, τις χρυσή τομής ε, μεταξύ αυτών των δύο ζητημάτων όλα αυτά γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε και ναι, περαιτέρω ανάπτυξη ακόμα και μέσα σε αυτό το τομέα. Κύριε Μπόρις, ο κύριος Μπόρις ανέφερε τα ίδια σημεία πάνω κάτω. Ελπίζω να απάντησα και τα δικά σας ερωτήματα. Ο κύριος Μπόρις όμως ρώτησε και για τα διευθυντικά ταμεία. Πώς ε, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε καλύτερα και πώς ε, μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Ισχύει αυτό που είπατε. Πράγματι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ε, ταμεία, τα διευθυντικά ταμεία σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά προγράμματα. Και από προσωπική πείρα, πριν από δεκαετίες, βεβαίως, στη δεκαετία του 80, στη Δανία είχαμε υψηλή ανεργία στους νέους και τότε ζητήσαμε πόρους από τα διευθυντικά ταμεία για να ε, εφαρμόσουμε ε, προγράμματα για την καταπολέμηση αυτής της ε, ανεργίας και έτσι δημιουργήσαμε πολλές θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι μαζί να σκεφτόμαστε και με διαφορετικούς τρόπους. Και έτσι ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε και νέε λύσει που ενδεχομένω δεν είχαμε σκεφτεί πριν. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και του δικού μου προγράμματος στον τομέα του πολιτισμού. Κυρία Κάμερβερτ, και εσείς αναφερθήκατε στο ρόλο των τεχνών και του πολιτισμού εν μέσω κρίσης και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τέχνες, να τις αξιοποιήσουμε για να δώσουμε ελπίδα στους πολίτες. Και αφετέρου ρωτήσατε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη βιομηχανία. Είναι σημαντικά στοιχεία για μένα. Ξέρουμε ότι η οικονομία διέρχεται κρίση, επομένως και ο πολιτισμός. Και τώρα για το πώς θα, θα... πρέπει να δούμε πώς θα ε, κάνουμε τον πολιτισμό έναν μοχλό ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν αυτή την ελπίδα που πρέπει να δημιουργηθεί και αφετέρου πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δημιουργική βιομηχανία είναι ένας από τους λίγους τομείς που, όπου αυτή τη στιγμή δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Από αυτές τις δύο λοιπόν οπτικές γωνίες θα πρέπει να εξετάσουμε τον πολιτισμό. Αφενός θα πρέπει να δημιουργεί ελπίδα και αφετέρου θα πρέπει να ε, συνεισφέρει στην, ε, στην ανάπτυξη της ε, βιομηχανίας. Μετά, πολλά ερωτήματα για τον αθλητισμό. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όσο το δυνατόν πληρέστερα. Κύριε Μπιλέτ, είπατε... Ρωτήσατε αν ε, θα ε, επιστήσουμε την προσοχή μας ε, στην, ε, στους, ε, στους managers, στους πράκτορες των ε, παικτών και εμάς μας εξέπληξε το μέγεθος αυτής της πρόκλησης και το ύψο ε, τη εγκληματική δραστηριότητα, το μέγεθο τη εγκληματική δραστηριότητα ε, στον αθλητισμό. Μιλούσαμε, είδαμε εκεί στήσιμο παιχνιδιών, ε, φαρμακοδιέγερση, ιδιαίτερα στου αθλητέ, αλλά όπω είπε και ο κύριο Μπελέτ, τη φαρμακοδιέγερση αυτή πρέπει να τη δούμε σε ευρύτερο πλαίσιο. Για παράδειγμα, στα γυμναστήρια. Όχι μόνο οι επαγγελματίε αθλητέ, Και εκεί βλέπουμε ότι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την ε, χρήση παράνομων ε, ουσιών. Αυτέ οι παράνομε ουσίε λοιπόν πλέον έχουν διαμορφώσει ένα μεγάλο, μια μεγάλη βιομηχανία, όπω και η βιομηχανία των ναρκωτικών. Στην Δανία έχουμε σχετικά θετικές εμπειρίες μέσω διαλόγου με αυτά τα γυμναστήρια και έτσι προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές ε, ε, πλαίσιο εγγύμνασης για τους ε, νέους μας ούτως ώστε να μην έρχονται αντιμέτωποι με την πώληση παράνομων ουσιών. Μία από αυτές τις δύο διασκέψεις ε, για τον αθλητισμό που ε, διοργανώνουμε στην ε, Κοπεχάγη αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι λοιπόν ένα θέμα που βεβαίως θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Ο κύριος Κόγη ανέφερε και τον προϋπολογισμό. Όπως και η συνάδελφός μου κυρία Αντορίνη, μπορώ να πω ότι είναι, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να, έχουμε, να είμαστε φιλόδοξοι σε πολιτικό επίπεδο. Αφετέρου όμως έχουμε και μια ιδιαίτερα δυσμενή πολιτική συγκυρία, οικονομική συγκυρία, συγγνώμη, και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι συζητήσεις για τον προπολογισμό ε, μένουν συνήθως ε, στον, στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών, όχι στο δικό μου τομέα. Βεβαίω όλα όσα αναφέρετε εγώ τα λαμβάνω υπόψη στο πρόγραμμά μου. Μετά, αναφέρθηκε κάποιος στο ζήτημα των ε, σλόγγαν στον αθλητισμό και της, ε, των συνθημάτων μάλλον στον αθλητισμό και την ε, παραπομπή στην σεξουαλική ταυτότητα των φιλάθλων. Εγώ έχω ε, συμμετάσχει σε διάφορες εκστρατείες ε, για αυτό το ζήτημα στα γήπεδα. Ε, αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αναλάβουμε και κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στην αλλά και πέραν τούτης, γιατί είναι σημαντικό να καταδείξουμε ότι αυτά τα συνθήματα μπορούν να έχουν και συνέπειες. Εμείς ως ηγέτες θα πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. Και τέλος... την κυρία Αναφερθήκατε στην, ε, στο, στη ψηφιακή ατζέντα, ψηφιακό πρόγραμμα. Ρωτήσατε πώς θα εξετάσουμε και θα χειριστούμε αυτές τις προκλήσεις των ψηφιακών κέντρων. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και πάλι το διαδίκτυο θεωρώ ότι προσφέρει πολλές ε, δυνατότητες ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου από την άλλη όμως θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα ε, πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Και για μένα αυτό είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία ισχυρής ε, βιομηχανίας στον τομέα της ε, πολιτιστικής δημιουργίας. Και πάλι λοιπόν αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Και τελευταίο ερώτημα των συναδέλφων. Ναι, δεν κατάλαβα καλά το ερώτημά σας. Μπορείτε να το επαναλάβετε. Δύο ερωτήματα για πώς θα ακολουθήσετε την κύρωση της σύμβασης της UNESCO. Είναι ένα ζήτημα που θέσατε στο έγγραφό σας και το άλλο αφορούσε τον πολιτιστικό τομέα ως τομέα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ποιε είναι οι προθέσει σα ε, σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ε, ε. Ναι, σε ό,τι αφορά την κύρωση της σύμβασης της UNESCO, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε επεξεργαστεί ήδη στη χώρα μου και είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Και είναι τμήμα της ε, πολιτικής της ε, Προεδρίας μας να δώσουμε μια διαπολιτιστική διάσταση στην πολιτική αυτή, όπως ε, αναφέρεται στο έγγραφό μας. Είναι και ένα στοιχείο λοιπόν του προγραμματός μας. που κινδυνεύει να χάσει <clears throat> την ε, προτεραιότητά του. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Προεδρία να υπογραμμίσει τη σημασία της πολιτιστικής πολυμορφίας, που είναι ακριβώς το αντικείμενο της σύμβασης αυτής της ε, UNESCO. Και νομίζω για τον πολιτιστικό τομέα σας έχω ήδη δώσει μια απάντηση. Πιστεύω ότι η δημιουργική, ο τομέας της δημιουργίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι ένας από τους λίγους τομείς που έχουν πραγματικά ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θετική ανάπτυξη δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και έχουμε πολλές δυνατότητες στον τομέα αυτό. Συγγνώμη, λέει ο κύριος ε, Λόκεργατ, για το θέμα της ε, συναπόφασης. Δεν νομίζω ότι το αναφέρατε το θέμα αυτό και για τα θέματα της ηθαγένειας. det som, det som øh, hvad hedder det, jeg selv er optaget af, og dermed også... Κοιτάξτε. Αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Προεδρία και εμένα προσωπικά είναι να δημιουργήσουμε μία ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα είναι κάτι που μπορεί να ξεκινήσει είτε από τις Βρυξέλλες είτε σε κάθε κράτος μέλος. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συνοχή και μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, ναι, χρειαζόμαστε τότε να δημιουργήσουμε μια ενιαία δημόσια σφαίρα. Ένα από τα στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν μια τέτοια δυναμική είναι αυτό το πρόγραμμα «Η Ευρώπη και τους πολίτες». Αυτό το πρόγραμμα και η οθέτησή του υπόκειται σε μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία. Ε, εγώ βεβαίως θέλω να πω ότι η συζήτηση ε, με την Επιτροπή σας ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, για τη διαμόρφωση αυτού του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας ως Προεδρία να έχουμε διάλογο μαζί σας και πιστεύω ότι ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο σας μεν για την ε, ενίσχυση δηλαδή της ευρωπαϊκής ε, κοινής γνώμης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων, μέσω των Εθνικών Μέσων Ενημέρωσης μπορούμε να καταστήσουμε πιο σοβαρή την όλη συζήτηση για την Ευρώπη. Και έτσι θα δώσουμε μια άλλη όθηση και στις εθνικές σχετικές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ίσως μπορώ να επανέλθω σε αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Λόκεγκαρτ και να τονίσω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται για αυτά τα προγράμματα η συναπόφαση. Το 2007 δεν ήταν έτσι, προηγουμένως δεν ήταν έτσι, πάντα προβλεπόταν η συναπόφαση σε τέτοια προγράμματα από τότε που υπάρχει ήδη από το 1992 η διαδικασία του 1992. Επομένως, προγράμματα όπως το Justitius που είναι πολύ σημαντικά για μας. Το ότι γίνεται μονάχα με διαδικασία σύμφωνης γνώμης και όχι με συναπόφαση, ότι αποφασίζονται πράγματα τα οποία δεν <clears throat> μπορούμε να τα επηρεάσουμε, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια τα, τις δυνατότητες που έχουμε σε επίπεδο νομικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα ζητήσουμε από την νομική μας υπηρεσία να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια στον τομέα αυτό. Δεν μπορώ να θεωρηθώ ότι αυτό είναι σωστό ως διαδικασία και ιδίως μετά από την εφαρμογή της ε, Συνθήκης Λισαβόνας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν κύριε Υπουργέ να κάνετε ό,τι μπορείτε για να υποστηρίξετε την αίτησή μας να υπάρξει η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας της συναπόφασης γιατί οι καλύτερες λύσεις βρίσκονται πάντα μαζί. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις απαντήσεις σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Ελπίζουμε λοιπόν στην Προεδρία κάθε μεγάλη επιτυχία στο έργο της. So, wir kommen jetzt zu Punkt 13. Σημείο 13 της ημερησίας διαταξής τώρα. Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών με, με γιώτα. Η κυρία Βερζιά έχει το λόγο. Je m'excuse. Φεύγει όλη η Δανία, λέει η πρόεδρο. Eh, Όλοι αυτοί που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν την επόμενη συζήτηση για την Ιθαγένεια, Σα παρακαλώ να βιαστείτε λιγάκι και να την κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φερισσιά, σα δίνω το λόγο. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών το 2013. Αυτό συνάδει και με τις ε, κατευθύνες γραμμές που έχουμε ήδη οθετήσει για την Ιθαγένεια. Το 2013 πράγματι θα είναι η 20η επέτειος της αποκατάστασης Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και ε, θα ακολουθηθεί από ανανέωση της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβει ισχυρό χαρακτήρα ε, να λαμβάνοντας υπόψη και τα πρώτα άρθρα της ε, Συνθήκης της για τη δημιουργία μιας ε, ισχυρής ένωσης ε, πάντα στο πλαίσιο ενός πνεύματος ανοιχτού και προσιτού στον πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διεξαγάγει ένα μεγάλο διάλογο με τους Ευρωπαίους πολίτες για να λάβει και τη δική τους άποψη για το πώς εκείνοι ε, βλέπουν ε, την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ιθαγένεια. Το λόγο μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση που μας ε, παρουσιάστηκε δεν είχε αυτό το πλαίσιο. Αρχικά για την νομική βάση. Η Επιτροπή στην πρότασή της ε, έλαβε μια ιδιαίτερα στενή έννοια του, ε, του ορισμού της αθαγένειας. Αλλά προτείνουμε όχι μόνο ένα ευρωπαϊκό έτο αθαγένειας, όπω είχε προταθεί στην έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτών, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό θα ε, μεταφράζεται πολύ καλά στην πρόταση που έχει γίνει. Αλλά υπάρχει χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και των ε, οργάνων, γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαιώματα, αλλά δεν τα γνωρίζουν. Και αυτό δεν είναι αναπαρκές κατά τη γνώμη μου. Ε, μιλάμε μόνο για, για τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και ουσιαστικά ε, θεωρούμε ότι μιλάμε μόνο για την άρση των εμποδίων ε, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, υπήρξε αντίστοιχη δράση το 2006 για την γενετικότητα και δεν ε, έχει νόημα να κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ιθαγένειας, ακόμα και δεν έχουν επιληθεί τα ζητήματα κινητικότητα. Μετά τις συζητήσεις που είχαμε τον εισηγητή και από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δεν συμφωνούμε με αυτή την ε, πολύπλοκη άποψη που υπάρχει για την ηθαγένεια. Θα πρέπει να επιλύσουμε λοιπόν αυτήν την κατάσταση, να λάβουμε υπόψη την εκπαιδευτική και πολιτιστική διάσταση της ηθαγένειας και πιο ευρέως να λαμβάνονται υπόψη και οι ε, λεγόμενες ε, η λεγόμενη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την συνθήκη Λισαβόνα, γιατί πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Δεν λέμε ότι πρέπει να ξαναγίνει η νομοδότηση του κυρίου Δεγάρτ, γιατί την υιοθετήσαμε σήμερα. Πρέπει να δούμε πώς η Ευρώπη μαζί με την Ευρώπη της Ιθαγένεια ε, ε, μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο. Πρόκειται για νομοθετική πρόταση και έχω υποβάλει περίπου 30 προτάσεις, ε, κυρίως για το προήμιο αρχικά, ε, που αφορούν τη σημασία της συμμετοχικής δημοκρατίας, της εκπαίδευσης ε, για ό,τι αφορά την ηθαγένεια, της αστικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, και εγώ αναφέρομαι σε μια έγκαιρη κατάρτιση ό,τι αφορά τις τα ευρωπαϊκά όργανα και διάφορα πολιτιστικά προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα για ε, την εκμάθηση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Μετά, για το ζήτημα της ε, ελεύθερης έκφρασης, ε, θα πρέπει να γίνει σεβαστή και η πολυγλωσσία. θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντα τον ρόλο των νέων, ε, των ε, διαφόρων ε, φορέων και το καθεξής. Δεν θα σας αναφέρω για τις 30 τροπολογίες, αλλά σε τρία σημεία. Πρώτον, για ό,τι αφορά την νομική βάση, η, η Επιτροπή ε, βάσισε την πρότασή της στο άρθρο 21 και μάλιστα μόλις στην παράγραφο 2. Και αυτό εξηγεί την πολύ στενή διάσταση που έχει λάβει πρόταση. Αναφερόμαστε στο άρθρο 20, πρώτη παράγραφος, ε, που καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Ακόμα λιγότερο όμως τα άρθρα 10 ε, και 11 και την συμμετοχική δημοκρατία και τις ε, σχέσεις των Ευρωπαϊκών Οργάνων με την κοινωνία των πολιτών. Δεν σας πρότεινα τροπολογίες με την στενή έννοια του όρου για την νομική βάση. Η πλειονότητα των τροπολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση οδεύουν αλλά έχουμε και τερμολογίε για τα άρθρα 165 και 166 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι αυτή η νομική βάση μπορεί να έχει συνέπειες, ε, ήδη ανέφερα κάποιες προηγουμένω για τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί σύμφωνα με την πρόταση, πρόταση της Επιτροπής να αλλάξουμε τη νομική βάση, βγαίνουμε από την διαδικασία συναπόφασης. Προτείνω να συνεργαστούμε στενά σε αυτό το ζήτημα με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που συμμερίζεται απόλυτα την άποψή μου. Προσθέτω ότι όσο περισσότερες τροποποιήσεις κάνουμε στην πρόταση της Επιτροπής, τόσο πιο δύσκολες θα είναι οι συζητήσεις με το Συμβούλιο και θα καθυστερήσουν, θα καθυστερήσει, καθυστερήσει συγγνώμη, η εφαρμογή της ε, πρότασης. Η Επιτροπή βεβαίω ε, θέλει να υιοθετηθεί η απόφαση πριν από τον Ιούνιο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα εργασία τη ε, με καλέ συνθήκε και για να διασφαλιστεί η επιτυχία του έτου Ευρωπαϊκή Σταγένεια 2013. Θα ήθελα επιμείνω στην αναγκαιότητα ε, των προγραμμάτων στο 8 και 17. Βεβαίω υπάρχει αυτή η συζήτηση για τα δημοσιονομικά και αυτό θα επιφέρει και τροποποίηση των προγραμμάτων. Νομίζω ότι αυτό το ευρωπαϊκό έτος ε, θα ε, είναι μια ευκαιρία να προβάλλουμε περαιτέρω τα προγράμματα που αφορούν ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. Τρίτο σημείο, ο προπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ευρωπαϊκής Ταγένειας, αν ακολουθήσουμε την πρόταση της Επιτροπής, θα έχει τον μικρότερο προπολογισμό που έχει ποτέ ε, δοθεί που έχει δοθεί ποτέ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. μικροσκοπικός προπολογισμός σε σχέση με ε, άλλα ευρωπαϊκά έτη. Η Επιτροπή επίσης λέει ότι και άλλα προγράμματα θα κινητοποιηθούν, όμως ε, εγώ είδα στο Ευρωπαϊκό Έτος ε, για τον εθελοντισμό και είδα τι συνέβη εκεί. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να μα πει ξεκάθαρα πώ βλέπει τα πράγματα, ποια θα είναι τα προγράμματα που ενδεχομένω θα κινητοποιηθούν. Περιμένω τι προτάσει τη Και βεβαίω θα τι ε, σημειώσω σε υποσημείωση ε, μέσα στο έγγραφο. Τώρα, με ή χωρί αλλαγή τη νομική βάση θα πρέπει να υπάρξει η ε, ε, σωσταθμιση τη διατύπωση για να λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή θαγένεια με όλε τι διαστάσει και η Επιτροπή των Περιφερειών και η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, συμφωνούμε με αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα όσα έχουν συμβεί και στους υπόλοιπους φορείς. Τέλος, πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Ευρωπαϊκής Θαγένειας μπορεί να είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να ανοίξουμε το διάλογο στα ζητήματα ηθαγένειας. Δυστυχώς, οι προτάσεις η πρόταση που μας έχει υποβληθεί δεν οδεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τέλος θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τον Σχιώδη, τους ε, συνεργάτες μας και τους συναδέλφους από την Επιτροπή. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Επιτροπής και συγκεκριμένα την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία που με βοήθησε πολύ. Και τέλος για την ε, καταληκτική ημερομηνία, αν με επιτρέπετε, πολύ σύντομα θα λήξει η προθεσμία. Έχετε μία εβδομάδα περίπου ε, για να υποβάλλετε προτάσεις τροπολογίας. Και αυτό γιατί αν θέλουμε να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες μας από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να δράσουμε ε, γρήγορα και προτείνω μια νέα ε, συνεδρίαση των σκεωδών στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βεζιά. Ο κύριος Σκούρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι με την εισηγήτρια βεβαίως στην εισηγήτρια που εξεφράστηκε για τον προπολογισμό. Φυσικά και δεν μπορούμε να αφιερώνουμε ένα ευρωπαϊκό έτος με όλα τα μηνύματα που συνεπάγεται, όπως είπε η Επίτροπος, με τόσο ελάχιστους πόρους. Τουλάχιστον εν μέρει ο προπολογισμό θα πρέπει να επαναξεταστεί. Ο δικός μου προβληματισμός πάντως σε σχέση με αυτά που μας είπε μόλις τώρα η συνάδελφος είναι ότι εσείς βασιστήκατε στην ιδέα του Ευρωπαϊκού Έτους της Ιθαγένειας, ενώ η Επίτροπος μας διευκρίνησε ότι μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών και τεκμηρίωσε ε, τη δική της αυτή επιλογή. Δεν ξέρω κατά πόσον οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να συγκρίνουν κατά πόσον υπάρχει κάποια, αν θέλετε, κάποιο πρόβλημα ε, και θα επηρεάσει και την τελική ε, υιοθέτηση της πρότασης. Θα θέλαμε να ακούσουμε με κάποια σαφήνεια και κατηγορηματικότητα από την Κομισιόν κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ όταν ε, είδα ότι δεν αναφέρθηκε το θέμα της Ιθαγένειας φαντάστηκα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό που έβγαλε το ψαλίδι Μπορεί τώρα να έχει κάνει μια διαφορετική άποψη, αλλά είναι γεγονό ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή ηθαγένεια, η Κομισιόν είναι παρούσα. Η κυρία Τιβέου, η κυρία Σότ, ποιο θα λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την συγκίτρια, την κυρία Βερσιά, για το εξαιρετικό της έργο σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν και για τις καρποφόρες επαφές που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σίγουρα η πολιτιστική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών. Και βλέπουμε σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια αρήκτο συνδέεται και με την κουλτούρα και με τα πολιτιστικά δικαιώματα και επομένως η Κομισιόν θέλει να χαιρετήσει τις πρωτοβουλίες αυτές που προέρχονται από την πολιτιστική πλατφόρμα και τα διάφορα προγράμματα δράσης στον χώρο αυτό. Αλλά για μας είναι σαφές ότι στους δύσκολους αυτούς καιρούς που μιλάμε για οικονομική κρίση ή όταν μιλάμε και για την κρίση εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα της λύσης και όχι του προβλήματος, όπως θεωρούν ορισμένοι. Και γι' αυτό η Κομισιόν έχει αναλάβει την ε, πρωτοβουλία να κάνει μια προσπάθεια να εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να κάνει, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, πώς μπορεί να δώσει λύσεις, πώς μπορεί να δώσει δυνατότητες και τι μπορεί να προσφέρει στους πολίτες σήμερα. και με συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τουλάχιστον για μας υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ των δικαιωμάτων της πολιτικής δέσμευσης και της συμμετοχής του πολίτη. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ηθαγένεια, γιατί αυτό ήταν από τα ερώτημα, ερωτήματα που τέθησαν, όταν ρωτάτε τους Ευρωπαίους πολίτες τι έρχεται στο μυαλό σας όταν μιλάμε για ηθαγένεια, σκέφτονται περισσότερο για την ελευθερία διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα από τα βασικά δικαιώματά τους. Και αυτό το οποίο έχει φανεί και στην έκθεση για την Ιθαγένεια και στα ψηφίσματα του <clears throat> Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι πολίτες δεν ξέρουν τα ποια είναι τα δικαιώματά τους, δεν ξέρουν ούτε καν ποιες είναι οι ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες για να ζήσουν καλύτερα τη ζωή τους και να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες που υπάρχουν για αυτούς ως Ευρωπαίους πολίτες. Για μας λοιπόν είναι και το θέμα να εντοπίσουμε ποια είναι τα εμπόδια στην ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια, αλλά και να αυξήσουμε και την επίγνωση των πολιτών για τα θέματα αυτά, να παροτρύνουμε συζητήσεις και μιλάμε και για δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, τα οποία δεν περιορίζουν μονάχα στην ελεύθερη διακίνηση και στην ελευθερία διαμονής και κατάστασης. Γιατί υπάρχουν πολλά δικαιώματα που είναι αλληλένδετα με αυτά τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν πραγματικά με την κοινωνική ασφάλιση, και τη δυνατότητα μεταφορά δικαιωμάτων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πολίτες στην καθημερινή του ζωή. Είπαμε επίση ότι ο στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτών ως ε, μια συνολική αιγίδα, μια συνολική ομπρέλα που θα καλύψει μια πληθώρα δραστηριοτήτων. Και για μας η το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών είναι πιο περιεκτική έννοια από το Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας. Γιατί έτσι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και τους νέους και αυτούς που είναι στα σχολεία. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε καμιά απολύτως ομάδα του πληθυσμού. Και όταν αναφέρεται επίσης η συγγήτρια στην έλλειψη αναφοράς στα νέα δικαιώματα που προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει απόλυτο δίκιο, γιατί μιλάμε και για τα άρθρα 10 και 11, αναφερόμαστε και για τη νέα πρωτοβουλία πολιτών και η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή εφέτος. Και υπάρχει και το ερώτημα για το είδος των άλλων προγραμματών που μπορεί να κινητοποιήσει κανείς και έχουμε ένα μακρό κατάλογο που μπορούμε πράγματι να εφαρμόσουμε μέσα στο έτος των πολιτών. Έχουμε προγράμματα για την ε, απασχόληση, <clears throat> για τους νέους οι οποίοι είναι σε κίνηση. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πολλά προγράμματα τα οποία θα συμμετάσχουν και άλλα εργαλεία της Κομισιόν στο έτος αυτών των πολιτών. Ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τους πολίτες της Ευρώπης και συζητάμε με όλους τους εταίρους μας και μέσα στην Κομισιόν και με τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών Υπάρχει λοιπόν μια ε, εντογενάστε συμμαχία, ένας συνασπισμός οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και αυτό θα βοηθήσει την Κομισιόν να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη διοργάνωση του έτους των πολιτών. Βασιζόμαστε φυσικά και στην αρρωγή των θεσμικών οργάνων και θα θέλαμε αυτό το έτος, το οποίο δεν είναι κάτι που επιβάλλεται εκ των άνω, όπως είπε η Κομισιόν, αυτά είναι θέματα που πρέπει να εκ των κάτω να προέλθουν τα θέματα συζήτησης. Ο στόχος είναι η συμμετοχή, ο ανοιχτός διάλογος και εν κατακλείδη έχει να κάνει με αυτά που αναμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να κινητοποιήσουμε όλους τους επλεκόμενους και στην κοινωνία των πολιτών και μέσα στα θεσμικά όργανα. Ετέθη ένα ερώτημα για τον προϋπολογισμό. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με τα προγράμματα που μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε μέσα στο έτος αυτό. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε όλες τις διαστάσεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση αποφασίσαμε να μην ζητήσουμε περισσότερα λεφτά. Γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης και υπάρχει επίκριση πολλές φορές ότι είναι πολύ δάπανα τα ευρωπαϊκά έτη και δεν παράγουν πάντα αποτελέσματα. Επομένως θα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία, ως πολιτικές, ως προγράμματα αυτά τα οποία έχουμε και μαζί με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα δράσουμε και ελπίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι επαρκής. Για μας είναι επαρκή τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να δημιουργήσουμε την απαραίτητη δομή για τη διοργάνωση αυτού του έτους γιατί βασιζόμαστε πολύ στη συνεργασία και στο συντονισμό με άλλους εταίρους. Οπότε η, η εστίασή μας, θέλω να το υπογραμμίσω, η εστίαση του έτους πολιτών και η εστίαση της πρότασής μας απορρέει από την έκθεση για τους πολίτες και το γεγονός ότι πολλές φορές οι πολίτες δεν έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω έλλειψης επίγνωσης αυτών, γνώσης και επίγνωσης αυτών των δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε ότι η εστίαση αυτή και η νομική βάση είναι η συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν και η ελπίδα μας είναι ότι με τις εξηγήσεις αυτές που σας έχω δώσει είναι κάτι το οποίο θα το κατανοήσετε και θα το αποδεχτείτε. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι, λέει η πρόεδρος. Θέλαμε να ξέρουμε γιατί ακολουθείτε, γιατί διαλέγετε ένα διαφορετικό τίτλο. Γιατί πήρατε την πρωτοβουλία να αλλάξετε τον τίτλο η Θαγένεια δεν έχει νομική βάση. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη νομική βάση στις συνθήκες. Γι' αυτό διαλέξαμε άρθρα που αναφέρονται στα πρόσθετα δικαιώματα που μπορούν να προσποριστούν οι πολίτες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν αυτών που τους παρέχει η εθνική τους ηθαγένεια ή η υπηκότητα. Και επομένως τα αρμόδια αυτά άρθρα της συνθήκης αναφέρονται στα δικαιώματα των πολιτών στους συγκεκριμένους τομείς. Ξέρω ότι κάποιος αναφέρθηκε στη συζήτηση στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό δεν επηρέασε την επιχειρηματολογία μας. Ευχαριστώ, όλοι οι πρόεδρες χωρίς μικρόφωνο. Θέλει συγγήτρια να πει κάτι. Ξέρουμε ότι η 1η Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, είναι πολύ σύντομα. Θα προσπαθήσουμε βέβαια στο βαθμό του δυνατού και του απαραίτητου να ε, βελτιώσουμε αυτή την έκθεση. Θα τα ξαναπούμε στο Στασβούργο. Σας ευχαριστώ για την εργασία σας και για να δούμε. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Σημείο 14. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για τα πορίσματα των συντονιστών. Α, επίσης, σας είχα ζητήσει για την επιστολή του κυρίου Ολιβάρης να την λάβετε υπόψη σας για τα θέματα των μελετών. Έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, κυρία Καμαρέβερτ. Λυπάμαι πολύ. για την προ... πρόταση μιας μελέτης για τους ε, πράκτορες των ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι αν περιοριστούμε μονάχα στο ποδόσφαιρο, είναι πολύ περιορισμένη αυτή η μελέτη. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να γίνει τόσο μεγάλος περιορισμός. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα τα οποία ενδεχομένω αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από ότι ε, το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό εγώ θα προτιμούσα να είναι πιο διασταλτική η διατύπωση και να μην περιλαμβάνει μόνο το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν σωστό. Γιατί έχουμε και το στίβο, έχουμε την κολύμβηση. Μπορούμε να το πούμε λοιπόν στην κυρία Ολιβάρες που είναι παρούσα εκεί ήδη ότι θα θέλαμε να έχουμε ένα ευρύτερο χώρο αθλητισμού. Εντάξει, δεν υπάρχουν άλλε αντιρρήσει. Έχουμε κλείσει και αυτό το σημείο. Έχουμε εγκρίνει τις αποφάσεις των συντονιστών. 29 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Όλη μέρα, πρωί και απόγευμα, στις 29 του μηνό. Σας ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία χθε και σήμερα και ελπίζουμε ότι έχουμε επιτύχει κάτι. Κλείνω λοιπόν την συνεδρία. Σας εύχομαι καλή όρεξη.